Mes chers collègues, nous allons ouvrir la séance, si vous voulez bien. Θα ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Ξεκινάμε με την υφέτηση της ημερήσία διαταξής μα. Τη θέλουμε και εγκεκριμένη αν δεν έχετε παρατηρήσεις και αντιρρήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια θλιβερή είδηση να σα ανακοινώσω. Όπως θα γνωρίζετε ήδη, ο συνάδελφός μας Γιένς Νίλσον απεβίωσε την περασμένη Τρίτη στις 12 του Μάρτη. Εξ ονόματος της Επιτροπής μας Μεταφορών και Τουρισμού και προσωπικά εξ ονόματός μου θα ήθελα να απευθύνω στην οικογένειά του και στους οικείους του όπως επίσης και στους συναδέλφους του καθώς και στην ομάδα των σοσιαλιστών τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και τους διασφαλίζουμε, τους εγγυόμεθα ότι είμαστε κοντά τους αυτή την δύσκολη στιγμή. Ήταν μια προσωπικότητα ο, ο Γιέντς που βρισκόταν μαζί μας από το 2011, ήρθε στην Επιτροπή μας το 2014 και ήταν μια προσωπικότητα που ήταν ευήκοη, ένα άνθρωπος ευήκοος. Ήταν πάντοτε ευχάριστο να ανταλλάσσει κανείς μαζί του απόψεις, ακόμα κι αν είχε κανείς διαφωνίες. Ήταν πάντα ανοιχτό στη συζήτηση και στο συμβασμό παραμένοντας ανυποχώρητος στις αρχές του. Ήταν ένας ε, πεπισμένος φιλευρωπαϊστής, στρατευμένος και περήφανος. Και εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι, όπως είδαμε κατά την ε, επίσκεψή μας στη Σουηδία τον περασμένο Ιούλη, στην πόλη που γνώριζε τόσο καλά, όπου ήταν ο Δήμαρχος μέχρι το 2009. Θα ήθελα εδώ εξ ονόματος όλων μας να αποτίσω φόρο τιμής στη δουλειά του και στους αγώνες του υπέρ των αγών, υπέρ της ισότητας ανδρών γυναικών κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης υπέρ των ατόμων με αναπηρία, υπέρ των συνθηκών εργασία των οδηγών. Και αυτοί οι αγώνες για την αξιοπρέπεια των ανδρών και των γυναικών παραμένουν στον πυρήνα της δουλειά μας. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω τις κόκκινες τυράντες του, το σήμα κατατεθέν κατατεθέντου που πάντοτε φορούσε με χάρη. Ήταν πάντοτε για μένα ένα μήνυμα και ένα σύμβολο απλότητας και προσβασιμότητας που ήταν περιβόητη. Θα παραμείνει μαζί μας αυτό στην Επιτροπή μας, όπως και ο ίδιος. Σας παρακαλώ συνάδελφοι να σηκωθούμε όλοι μαζί και να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του συναδέλφου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνήθι μας Ισμαήλ του εξ ονόματος των Σοσχριστών Ισμάλερ έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για αυτό το φόρο τιμή στη μνήμη του συναδέλφου Γέντς Νίλσον. Πιστεύω ότι αυτές οι στιγμές είναι όντω πολύ θλιβερές για όλους μας, για όλη την πολιτική μας ομάδα και όλους τους συναδέλφους του συναδέλφου Νίλσον που ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένας πολύ φιλικός συνάδελφος και δεν ξέρω αν οφείλεται στο σκανδιναβικό του ταπεραμέντο, αλλά πάντοτε αναζητούσε ισορροπίες και συμβασμούς μεταξύ των θέσεων μας. Ήταν ενεργό σε διάφορους τομείς, κυρίως υπέρ των αδυνάτων. Πάντοτε θα τον τιμόμαστε λοιπόν. Και για το χαρακτήρα του θα ήθελα να πω ότι ποτέ, μάλλον πολύ σπάνια στην πολιτική συναντά κανείς ένα τόσο φιλικό, τόσο ισορροπημένο άνθρωπο και στην ομάδα μας των σοσιαλιστών είχε διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στα θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών, θέματα που του ήταν προσφυλή και που είχε προσπίσει εδώ και στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Μεταφορών, με τρόπο παραδειγματικό. Για μας είναι μια μεγάλη απώλεια. Θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ο Γέντς Νίλσον ήταν ένα φανταστικό άτομο εύχομαι στους οικείους και στην οικογένειά του κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και απευθύνω, τους απευθύνω στα τα θερμά μας συλληπιτήρια εκ μέρους των σοσιαλιστών, εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας μας. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο και με βέβαιος ότι πολλοί συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μαζί μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την βοηθό του την Πέτρα που του συμπαραστάθηκε σε πολιτικό τεχνικό επίπεδο. Είχαμε φτιάξει μια καλή ομάδα με τον Γέλντς και ευχόμαστε και πάλι στους οικείους του καλό κουράγιο, καλή δύναμη και ευχαριστώ μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Ισμαέλ Σας ευχαριστώ πήρατε το λόγο εκ μέρους των σοσιαλιστών. Και θα ήθελα να πω προς τους ε, βοηθούς του κυρίου Γιάννη ότι η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντα ανοιχτή ό,τι και αν συμβεί. Ξέρω ότι είναι μια θλιβερή στιγμή, συνάδελφοι, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε και εμείς τη μάχη μας και σήμερα θα εργαστούμε στη μνήμη του και θα συνεχίσουμε με την μέσια μας διάταξη. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε προηγουμένως όλους σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη μέση διάταξή μας και θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λιμπεράτσκι Γεια σας κύριε Λιμπεράσκη. Τι κάνατε, είστε καλά, λέει πρόεδρος. Θα μας παρουσιάσετε το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σε διεροδρομικών μεταφορών. Συνάδελφοι, υπενθυμίζω ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αφορά εκατομμύρια συμπολίτες μας και κυρίως αφορά εκατομμύρια συμπολίτε μας όσον αφορά τις ελλείψεις ενός μεταφορικού μέσου όπως οι συνδρομικές μεταφορές που διευκολύνουν πολύ την καθημερινή μας ζωή. Οπότε κύριε Λιμπεράσκη θα δώσω το λόγο σε εσά, αλλά και στους ε, σκέδους συζητητής και στους αδέλφους που το επιθυμούν για να μιλήσουν. Θα δώσω επίσης και στον κύριο Κουλόν από την ε, ε, και τον λόγο. Καλημέρα και ο Κουλάν, είστε καλά. Για να μάθουμε την άποψη και την γνώμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ε, και Κοινωνικής Επιτροπής και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Κύριε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλή εισαγωγή σας είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εισηγητής για αυτό το ζήτημα και κάνω ό,τι μπορώ για να κάνω στην καλύτερη δουλειά. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο στοιχεία. Πρόθεσή μου είναι να συνδυάσω ε, τις δύο πλευρές του ζητήματος και τους παρούχους υπηρεσιών και τους ε, πελάτες, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Πρέπει και να προσελκύσουμε ε, πελάτες, ιδάλλως δεν θα υπάρχει και ζήτηση. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε την ε, ισορροπία. Η βασική πράξη ήταν του 1991. Εδώ και πολλά χρόνια λοιπόν έχει αρχίσει η θέσπιση ενός ε, πλαισίου πλέον απαιτούνται ορισμένε τροποποιήσει ρυθμιστικέ και κανονιστικέ ε, με βάση τι εξελίξει στον κλάδο. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν σημαντικέ αλλαγέ και διαφορέ μεταξύ τμήματων και περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να καλύψουμε, να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ τους. Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου είναι καλό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και καλύτερο. Θα πρέπει να διαμορφώσει τις συνθήκες ε, μονίμου βελτίωσης για τον κλάδο. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται και σε ό,τι αφορά την προστασία των επιβατών πρέπει ο επιβάτης να νιώθει προστατευμένος και ασφαλής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η διασύνδεση ε, μεταξύ των ε, παρόχων υπηρεσιών και των επιβατών. Η ιδιαίτερη μνήμη γίνεται για, για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Κάναμε πολλές ε, συζητήσεις από αυτού Νομίζω ότι έχω λάβει γνώση της κατάστασης και νομίζω ότι την έχω ε, απεικονίσει με τον κατάλληλο τρόπο στην έκθεσή μου. Το σημαντικό είναι ε, οι υπηρεσίες αυτές να είναι προσιτές και από οικονομικής ε, πλευράς και από πλευράς δυνατότητας φυσικής πρόσβασης και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα συνδρομικών μεταφορών με έναν ανοιχτό χώρο συνδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, θέλουμε να δημιουργηθεί ένα ίσο πεδίο ανταγωνισμού και σε σχέση με άλλους ε, τρόπους ε, μεταφορών. Πρέπει ο ανταγωνισμός να είναι δίκαιος. Με περιορισμένη γραφειοκρατία για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Το σχέδιο έκθεσης προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με 21 Συναδέλφου 21 διαφορετικά μέρη και από τον συνάδελφο Αλεξάνδρ Φόχτ ε, με πάνω από 40 συνεδριάσει και κάναμε και μία μικρή ακρόαση το Φεβρουάριο. Από πλευρά μου έχω καταθέσει 55 τροπολογίες που δημοσιεύθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και εν μέρη συζητήθηκαν στις 6 Μαρτίου στην ομάδα εργασίας μεταφορών των σοσιαλιστών. Θα λοιπόν να είναι προσιτές προς όλους τους ε, πολίτες ε, οι υπηρεσίες αυτές και πιο συγκεκριμένα και προς τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα να περιορίσουμε την άνηση μεταχείριση των σιδηροδρόμων σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς και να βελτιώσουμε την διαθεσιμότητα των εισιτηρίων, λάμβανοντα υπόψη και ε, λύσει με βάση τον κλάδο που ήδη έχουν υιοθετηθεί. Θέλω να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα ε, της ε, πολυτροπική και ενδοτροπικής προσέγγιση σε ό,τι αφορά τους αεροδρόμους, ούτω ώστε να ικανοποιούνται και οι πελάτες. Για τι εξαιρεσει τώρα. Το πεδίο εφαρμογής προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις που προτείνω να διατηρήσουμε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Οι εξαιρέσεις αφορούν τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 13. Βέβαια, ουσιαστικά πρόκειται για 11 κράτη-μέλη, γιατί οι άλλα δύο δεν έχουν σιδηροδρόμο. Γιατί μέχρι το 2024 γιατί αυτό το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μας δίνει δυνατότητα ε, αναβάθμιση των ε, υποδομών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2024. Γι' αυτό θέτουμε αυτό το χρονικό όριο. Για να αρχίσει δηλαδή η θέση σε ισχύ ε, και η εφαρμογή αυτών ε, των κανόνων σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών. Μετά τροπολογία 36, 37, 24 και στα παραρτήματα έχω βάλει κάποιες ε, προκειμένου να έχουμε ενιαία θηρίδα για τους ε, επιβάτες και για να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις με το τρίτο πακέτο. Γιατί είχα τη δυνατότητα να εργαστώ μαζί σας ε, ε, σχετικά με τη δέσμη σιδηροδρομικών μέτρων. Με την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων όμως, γιατί μπορούν να θεωρηθούν αντίφαση. η βελτίωση της προσβασιμότητα και της συνδρομή προ του επιβάτες περιορισμένη κινητικότητας. Ο εισηγητή θεωρεί ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δεν αντικατοπτρίζει ε, τις ανάγκες, γι' αυτό θα πρέπει όλο το συνδρομικό ε, σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προσβάσιμο ε, εντός 24 ωρών για όλα τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διατηρήσει το χρονικό όριο των 48 ώρων. Αυτό καλύπτεται την τροπολογία 44. Ήδη σήμερα οι μεγάλοι σταθμοί ε, διασφαλίζουν την πρόσβαση με ή χωρίς πρώτερη ειδοποίηση κάτω από τις 24 ώρες. Θα πρέπει η συνδρομή να παρέχεται δωρεάν. όπως αναφέρω και στις τροπολογίες 40 44. Επιπλέον, οι αρχές επιβολής του νόμου στο εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ε, διεξαγάγουν ε, ελέγχους ε, στα συστήματα των σταθμών για να εντοπίζουν ανεπαρκείς υπηρεσίες ή υποδομές στους συνδρομικούς σταθμούς. Όπως και να έχει να σαφές ότι αν επιβάλλουμε υπερβολικά αυστηρούς κανόνες και στους μικρούς δεύτερο δευτερογενεί, ίσως σημασία δηλαδή, σταθμούς, τότε αυτό θα είναι αρνητικό για μέρο ε, τουλάχιστον του συνδρομικού συστήματο. Προσβασιμότητα των ε, εισιτηρίων. Η διαθεσιμότητα είναι σημαντικό στοιχείο για την αύξηση της ελκυστικότητας ε, των σιδηροδρόμων, αυτό που ανέφερα και στην αρχή. Θεωρώ όμως ότι δεν αναπόκειται στο νομοθέτη να επιβάλλει υπερχρεωτική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα σε ένα πλαίσιο ανοίγματο της αγοράς. Ο σιδηροδρομός θα πρέπει ε, να τύχει της ίδιας μεταχείρισης με τους άλλους τρόπους μεταφοράς και να, θα πρέπει να του δοθούν οι απαραίτητες ευκαιρίες για να αναπτύξει αυτές τις λύσεις από μόνος του. Από αυτή την άποψη η οδηγία 2016 κάθετος 2370 13α άρθρο προβλέπει ότι ο κλάδος των συνδυοδρόμων θα πρέπει να βρει πρωτοβουλίες της αγοράς μέχρι το 2022. Εδώ σήμερα έχουμε το Full Service Model, το οποίο έχει αναπτυχθεί από ε, συγκεκριμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, 17 τον αριθμό, και θέλουμε να ενθαρρύνουμε και άλλες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα, όπως το Trainline, Silver Rail και ούτε καθεξής, για να παρέχουν διασυνοριακές ε, μεταφορές και μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. Μετά, όταν, έχουμε, όταν κάποιος χάνει την ανταπόκρισή του εδώ και κανένα δύο χρόνια 14 επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει εμπορικής συμφωνίας διασφαλίζουν ε, τα ταξίδια σε περίπτωση διαταρχής ε, του ταξιδιού και σε αυτό συμμετέχουν ε, όταν έχουμε ένα ταξίδι με διαφορετικές επιχειρήσεις, διαφορετικές εταιρείες. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν αυτά τα συστήματα. Όλα αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι ο σιδηροδρομικός κλάδος ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Κάποιες φορές και από μόνο του ο κλάδο ε, αναλαμβάνει δράση. Γι' αυτό προτείνω να τηρήσουμε την προθεσμία του, της τέταρτης δέσμης για το σιδηρόδρομο. Πέραν της διαθεσιμότητας, των εστηρίων. Θα πρέπει πάντα ο επιβάτης να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του όταν ένα ε, συνδρομικό ταξίδι ε, περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατηγορίες ναύλων. Ανατέρα βία. Αυτό έχει συστηθεί επί μακρόν. Πρόταση είναι να συμπεριληφθεί εξαιτία του ανταγωνισμού μεταξύ του σιδηροδρόμου και των αερογραμμών. Για παράδειγμα, έχουμε μεγάλες πόλει και συνδέσεις, ε, για παράδειγμα, μεταξύ Βρυξελών, Παρισίων ή Βρυξελών, ε, Λονδίνου, όπου υπάρχει ανταγωνισμός ε, μεταξύ του σιδηροδρόμου και των αεροπορικών αερογραμμών. Ε, προς το παρόν ο σιδηρόδρομο δεν προβλέπει ανωτέρα βία, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν και τέτοιε περιπτώσει, όπω και στην περίπτωση τρομοκρατία. Θεωρώ λοιπόν ότι η ανωτέρα βία θα μπορεί να βασιστεί ε, στου θεσπισμένου ε, κανόνε ανωτέρα βία με βάση την τροπολογία 34. Από την πλευρά των ε, επιβατών των σιδηροδρόμων, θεωρώ ότι ο επιβάτης δεν ε, περιμένει απαραίτητα αποζημίωση από τον πάροχο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτεί και περιμένει μάλλον ο επιβάτης συνδρομή, η οποία παρέχεται με βάση το σχέδιο της έκθεσης. Περαιτέρω τροποποιήσει στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένες αλλαγές που έχει προτείνει η Κομισιόν δυστυχώς είναι επιζήμιας προς το μέλλον ε, των σιδηροδρομικών γραμμών. Και κάποιες φορές, μάλιστα, δεν ακολουθούν και τους κανόνες της κοινή λογικής. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το άρθρο 16, σημείο 2, που λέει ότι η συνδρομική επιχείρηση θα πρέπει να βρίσκει νέο δρομολόγιο όταν υπάρχει πρόβλημα ο εισηγητής θεωρεί ότι το τρέχον 16 καλύπτει τις ε, απαραίτητες επιλογές. Δίνει τη δυνατότητα μεταξύ πλήρους αποζημίωσης του ναύλου, ε, rerouting, δηλαδή ε, να συνεχίσει ο επιβάτης το ταξίδι του το δυνατόν ή να βρεθεί νέα λύση, νέο ταξίδι, όποτε αυτό βολεύει τον επιβάτη. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες. Τώρα για να δώσουμε αποζημίωση για τα εποχιακά ε, εισιτήρια. Δεν είμαστε πεισμένοι για τεχνική σκοπιμότητα αυτού του μέτρου που θα επιφέρει και επιπλέον διοικητικό άχθος. Γι' αυτό έχουμε τροπολογία 32. Τέλος, η κακή κατάσταση των υποδομών σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν ε, οφείλεται ε, στην αμέλεια των ε, σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, αλλά προκύπτουν συχνά από τις εθνικές πολιτικές στον των μεταφορών που δεν επενδύουν στο σιδηρόδρομο. Όμω, έχουμε δυνατότητα να καλύψουμε αυτό το χάσμα με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τέλος, ε, μελλοντικέ κινήσεις. Υπάρχουν προτάσεις ε, αναστολής ή αναβολής ορισμένων ε, προτάσεων. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε εμεί. Όπως και να έχει, προβλέπουμε Προθεσμία κατάρτιση τροπολογιών 27 Μαρτίου 2018 στις 11 το πρωί. Η επόμενη συνάντηση των σχεδόν 17 Απριλίου θα λάβει χώρα. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται τον Ιούνιο του 2018. αν πραγματικά θέλουμε να ολοκληρωθεί η εξέταση της πρότασης ε, μέχρι το τέλος της θητείας, θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό το ε, χρονοδιάγραμμα, να μην ξεφύγουμε από αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας και για την πολύ καλή εισαγωγή, κυρία Πρόεδρε. Euh, σας ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Ξεπεράσατε κάπως το ρόλο σας του εισηγητού διότι βεβαίως ε, το χρονοδιάγραμμα για τα παραπέρα βήματα θα το δίνω εγώ. Αλλά σας συγχωρώ. Ας δούμε λοιπόν. Αρχίζει η και θα αρχίσω με εσάς κύριε Μισελιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και χαίρετε σε όλες και όλους ο Αντιπρόεδρος κ. Λιμπεράσκη, τον ευχαριστώ για την έκθεση και για τις πρώτες τροπολογίες για την τροποποίηση του κανονισμού για τις ιδρυοδομικές μεταφορές. Ελπίζω να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, να προχωρήσουμε γρήγορα στην ουσία για τους ε, χρήστες των σιδηροδρόμων, αλλά έχω και ορισμένε αποκλήσει από τις απόψεις του εισηγητού πρέπει να μπει ο κανονισμός αυτός στην ε, μεγάλη αναθεώρηση των σιδηροδρόμων. Να νομοθετηθούν τα δικαιώματα των επιβατών, διότι αυτά πάνε χέρι με χέρι με το άνοιγμα των αγορών των σιδηροδρόμων. Δηλαδή, επιτυχημένος ανταγωνισμός πρέπει να βασίζεται και σε εναρμονισμένα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων επιβατών. Έτσι μόνο θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επιβατών απέναντι στους σιδηροδρόμους, των χρηστών δηλαδή. Και θα προωθήσουμε και την ανταγωνιστικότητα και τις διατροπικές μεταφορές. Αποτελεσματικότητα. Επίσης, χρειάζονται μέτρα να εφαρμοστεί το κείμενο στο σύνολό του και χωρίς ε, εξαιρέσεις αποκλήσεις από το 2019. Οι εθνικές αγορές που θα ανοίξουν στην, στον ανταγωνισμό θα λειτουργούν στην ίδια βάση και με ένα ελάχιστο όριο ίσων κανόνων. Για τους περιφερειακούς υδροδρόμους αυτοί θα ανοίξουν στον ανταγωνισμό το αργότερο το 2019. Διότι να υποφεληθούν όμως το 90% των εκβατών αυτό μου φαίνεται απίθανο. Μετά από την έγκριση του πρώτου κανονισμού μόνο τέσσερις χώρες μέλη τον σέβονται και μπράβο τους. Αυτό είναι θετικό για τον φορολογούμενο και για τον χρήση του σιδεδρόμου. Για τους υπολείπους όμως δεν σέβονται τους επιβάτες τους. Δεύτερο. Να διευκολυνθεί ο επιβάτης και να είναι ασφαλής στο ταξίδι του. Όποιος και αν είναι ο λόγος για τον οποίο ενδεχομένως χάνει το τρένο του, να του δίνουν αυτομάτως θέση στο επόμενο τρένο, όποιος και αν είναι ο operator του τρένου αυτού. Αυτό πρέπει να, να συμβαίνει για όλα των, ειδών τα εισιτήρια και να λυθούν υπόψη οι ανάγκες των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες και αναπήρων, διότι μιλούμε εδώ για 80 εκατομμύρια πρόσωπα. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν στοχεύσουμε τις προσπάθειές μας στην ε, προστασία της καθημερινής κινητικότητας. Να μπορεί ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως της προσωπικής τους κατάστασης. Δέχομαι λοιπόν τις προτάσεις του εισηγητού για να μειωθεί η προειδοποίηση 24 ώρες για την παροχή ε, βοήθειας στον επιβάτη και αναλόγως βέβαια με την πυκνότητα των σταθμών. Τέλος, να επανεξεταστεί το ζήτημα των ε, αποζημιώσεων για οποιαδήποτε καθυστέρηση και να προσαρμοστεί στις πραγματικότητες του σιδηροδρόμου και να μειωθεί το, ε, κατόφλι, το επίπεδο δηλαδή από το οποίο και μετά χορηγείται η αποζημίωση σε 30 λεπτά. Έτσι θα ενθαρρύνουμε περισσότερους ε, ανθρώπους να μην παίρνουν το αυτοκίνητο για τις μικρές διαδρομές. Χρειάζονται λοιπόν κίνητρα και αντικίνητρα. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι υπεύθυνε Βέβαια, όταν υπάρξει ανταγωνισμό, η λογική του ανταγωνισμού θα τι αναγκάσει να είναι πιο αποδοτικέ και να προσφέρουν καλύτερο ε, καλύτερες υπηρεσίες στον επιβάτη σύμφωνα και βέβαια και με το ύψο των φόρων που καταβάλει και είναι, έχει ε, το δικαίωμα να τα ζητεί αυτά τα πράγματα. Θα συνεργαστούμε για να κάνουμε πραγματικότητα αυτό, αυτή την επανάσταση στους σιδηροδρόμου. Επανάσταση των επιβατών. Ευχαριστώ κύριε Μιζελή. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θερμά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Δεν είμαι εγώ σκιώδη εισηγητρία για το θέμα αυτό. Αλλά πάντως ε, μπορώ να σας πω τι σκεπτεί η ομάδα μας. Νομίζω ότι ο εισηγητής εξήγησε με σύντομο τρόπο όλους τους τομείς στους οποίους συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μια και είμαι Ευρωβουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουμε ήδη ξεπεράσει πολλά από τα ελάχιστα στάνταρτ τα οποία περιλαμβάνει η υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Να διασφαλίζουμε δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν υποχωρήσει. Πρώτο λοιπόν, PRM, δηλαδή ε, επιβάτε με περιορισμένη κινητικότητα. Εδώ χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη ανεξαρτήτως του ότι κάποια φορά είναι ε, δύσκολο διότι υπάρχουν πολλοί παλαιοί σταθμοί σε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει να είναι δυνατόν όχι μόνο στους σταθμούς αλλά να τη βοήθεια στα, στους επιβάτες αυτούς και μέσα στους σειρμούς είτε με ράμπες είτε αλλιώς. Πολύ σωστά λοιπόν ανάγεται το θέμα αυτό σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της αναθεώρησης του κανονισμού για το through ticketing, για το εισιτήριο για όλη τη διαδρομή. Από την πρώτη μου εντολή ήδη 2002-2003 μας απασχολούσε το θέμα αυτό. Δεν έχουμε προχωρήσει πολύ και νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει ζήτημα κλειδί. Θέλουμε οι άνθρωποι να μπορούν να κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις με αυτά τα γρήγορα τρένα και είναι πολύ απογοητευτικό όταν από τη μια χώρα στην άλλη είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να έχουν ε, εισιτήριο για ολόκληρη τη διαδρομή. Χαίρομαι λοιπόν που τονίζεται το σημείο αυτό, κύριε Σιγητά, διότι νομίζω ότι πολλοί από του operators, πολλέ από τι επιχειρήσει δηλαδή, πρέπει να κάνουν προσπάθειε εκεί. Σε ό,τι αφορά τι εξαιρέσει. Ε, σύμφωνοι για το 2024, πολύ λογικό να συνεχίσει να ισχύει η ημερομηνία αυτή, η χρονολογία αυτή. Τέλος, μιλήσατε για την ανωτέρα βία. Σωστά είπατε ότι η ανωτέρα βία, αν το σκεφτεί κανείς καλά, ισχύει για όλα τα είδη μεταφορών. Είτε πρόκειται για λεωφορείο, είτε πρόκειται για πλοίο, είτε πρόκειται για αεροπλάνο. Χρειάζεται λοιπόν να ορισμένα πράγματα που ξεφεύγουν από τον έλεγχο των εταιριών. Αλλά θα πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιείται η ίδια ορολογία εμείς λέμε στις ε, αερογραμμές duty of care, δηλαδή ε, ανάγκη της δέουσας επιμέλειας. Και θα πρέπει οι πελάτες, οι επιβάτες δηλαδή να είναι ενημερωμένοι και όπου υπάρχει υποχρεωτικό καθήκον δέουσας επιμέλειας πρέπει τα πρόσφατα να βοηθούν το δυνατόν συντομότερο και ιδίω να μπορούν να φεύγουν και να συνεχίζουν το ταξίδι τους όταν για παράδειγμα υπάρχουν δυσμενεί μετεωρολογικέ συνθήκες ή όταν υπάρχουν απεργίε κλπ. Νομίζω ότι είναι, προσω... Ε, ε, ε, ισορροπημένη η προσέγγιση του εισηγητού. Εμείς σας υποστηρίζουμε ως ομάδα των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών και σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ κυρία Φώστερα. Ο κύριος Βαν Χούλτενβερκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι παρόν σήμερα ο σκιώδης ηγητής μας. Γι' αυτό θα σας πω λίγο αυτά που θα ήθελε. Ως φιλελεύθεροι λαμβάνουμε υπόψη το σχέδιο του ηγητού. Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι ο νέος κανονισμός στοχεύει πραγματικά στα συμφέροντα του επιβάτη, που ο επιβάτης θα πρέπει να είναι στην καρδιά των ρυθμίσεων, διότι ζητούμε εναρμόνιση ή υψηλά επίπεδα ε, ε, ελάχιστων κοινών κανόνων για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. δυστυχώ όμω ο ε, εισηγητή αποδυναμώνει ορισμένε ρυθμίσει που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή εξαιρέσει, χαμηλά επίπεδα ορισμένων υπηρεσιών και ούτω Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι λυπηρό, διότι ο κανονισμός απεδείχθη ο ισχύων δηλαδή ότι είναι ανεπαρκής από την άποψη προστασία των επιβατών. Και αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι αποδεκτό. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες και για το through ticketing. Θα πρέπει δηλαδή οι πελάτες, οι επιβάτες να έχουν τι δυνατότητες να επιλέγουν όλες τις ε, επιλογές ώστε να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό ανεξαρτήτως ας πούμε καθυστερήσεων ή εσφαλμένων διασυνδέσεων κλπ. Άρα Όλα αυτά είναι αναγκαία για να υπάρξει ισότιμος ανταγωνισμός και να γίνει ο σιδηρόδρομος πιο ελκυστικός και να εξασφαλιστεί η ανάπτυξή του και να αυξάνει και ο αριθμός των επιβατών. Είμαι σκιώδης για την γνωμοδότηση της ΙΜΚΟ και σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού. Στην έκθεση ΙΜΚΟ θα βάλουμε τον καταναλωτή ασφαλώς πρώτο και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία και για τη δική σας Επιτροπή, Επιτροπή Μεταφορών, Τραν, πιο συγκεκριμένα. Για να τον υποστηρίξει η ομάδα Άλντε θα πρέπει ο εισηγητής να δείξει διάθεση να ξανασυζητήσει τα πράγματα που ανέφερα προηγουμένω. Σας ευχαριστώ και τον ευχαριστώ και για την προσοχή του. Ευχαριστώ κύριε Βαν Μέντενμπερκ, ο κύριος Κάμερ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή κ. Λιμπεράτσκι και αναμένω καλή συνεργασία μαζί του και για το μέλλον, διότι και οι δύο είμαστε υπέρ του σιδηροδρόμου. Είναι κρίμα που δέκα χρόνια από τότε που ψηφίστηκε η σχετική νομοθεσία που λειτουργεί καλά σε ορισμένε χώρε μέλη, καλούμεθα τώρα να φτιάξουμε νέα νομοθεσία. Διότι μόνο τέσσερις χώρες μέλη μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο. Εκεί όμως μετέφερε στο εθνικό δίκαιο λειτουργήσε καλά το σύστημα. Και γι' αυτό δεν υπάρχει αφορμή, δεν υπάρχει λόγος να αποδυναμωθεί η νομοθεσία. Καλύτερα να διδαχθούμε από τα ασφάλματα που έχουν γίνει για να τα βελτιώσουμε. Να μην επιτρέψουμε εξαιρέσει, διότι τότε οι χώρες μέλη μπορούν να πούν «Α, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν μας ενδιαφέρει δε». Τώρα, έχουμε σε ορισμένα επιμέρου θέματα. Για παράδειγμα, ανωτέρα βία. Και ρωτώ, γιατί να εισαχθεί τώρα η ανωτέρα βία που δεν υπήρχε πριν και δεν είχε αποτελέσει και πρόβλημα. Νομίζω σε 15 χρόνια, σε 15 χρόνια από την Ομοσπονδία Επιβατών χρειάστηκε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να επενδυθούν ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την ανωτέρα βία. Γιατί τα χρήματα αυτά να μην πάνε καλύτερα υπέρ των επιβατών. Γνωρίζουμε και από τις αερογραμμές ότι η ανωτέρα βία έχει οδηγήσει σε σωρία δικών που τελικώς δεν οδήγησαν πουθενά και ο κόσμος τελικώς τα εγκατέλειψε. Ας κάνουμε μια ασφάλιση. Κοστίζει πολύ λίγο. Υπάρχει όμως. Και οι ιδιώτες έχουν λοιπόν, ως ιδιώτες εννοώ, ασφάλιση για ανώτερη βία. Για παράδειγμα, άμα πιάσει φωτιά το σπίτι τους. Ας κάνει το ίδιο και η ε, σιδηροδρομική εταιρεία. Άλλο, το through ticketing, ότι δεν έχει ακόμα φτάσει η είδηση αυτή μέχρι του ιδεοδρόμου, ότι δεν έχουν αναλάβει η ίδια πρωτοβουλία. Με τον τρόπο αυτό όμω υποσκάπτουν τον ανταγωνισμό, υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητά του απέναντι στου άλλου τρόπου μεταφορών. Θα πρέπει τουλάχιστον για ολόκληρη την Ευρώπη να έχω στη διάθεσή μου ως επιβάτης όλε τι πληροφορίε, Πότε φεύγουν τα τρένα, από πού, καθώ και τι τιμέ. Αυτά τα βλέπουμε ήδη στι περιφερειακές συνδέσει και στο Βερολίνο υπάρχουν πάνω από 30 λεωφοριακές γραμμές οι οποίες συνεννοούνται μεταξύ τους και προσφέρουν την υπηρεσία αυτή. Και εν τέλει ο επιβάτης δεν ενδιαφέρεται ποιος ακριβώς θα το μεταφέρει, αρκεί να πάει στον τόπο προορισμού του. Κάτι που ε, επίσης είναι σημαντικό είναι βεβαίως οι επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα. 48 ώρες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 48 ώρες δηλαδή θα πρέπει να λέει ο άνθρωπος που έχει ανάγκη το αναπηρικό κάθισμα, 48 ώρες, ότι θα πάω στον τάδε σταθμό και χρειάζομαι κάποια βοήθεια. Αυτά είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός βεβαίως ψηφιακής εποχής. Και εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε. Πού λειτουργούν τα πράγματα αυτά, ορίστε, στις κάτω χώρες λειτουργούν. Μία ώρα πριν, μία ώρα πριν πετυχαίνει. Μπορεί, έχει την υποστήριξη ο άνθρωπος που χρειάζεται. Και αφού πετυχαίνει στις κάτω χώρες, γιατί δεν μπορεί να πετύχει και στη Γαλλία ή στη Γερμανία αυτή η παρα, παλαβή ιδέα της Κομισιόν, δηλαδή 48 ώρες, ενώ έχουν το θετικό, το παράδειγμα μάλλον των ε, κάτω χωρών. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Κάτι άλλο το οποίο με ενδιαφέρει βέβαια πάρα πολύ είναι η δυνατότητα να πάρει κανείς το ποδήλατο μαζί. Και αυτό το είχαμε αποφασίσει προ δεκαετίας. Να είναι δυνατό να παίρνει κανείς το ποδήλατο μαζί σε όλα τα τρένα μεγάλης ταχύτητας. Μετά από πιέσεις της γερμανικής κυβέρνησης και των γερμανικών σιδηροδρόμων μπήκε και μια φρασούλα που λέει εάν αυτό είναι εύκολο και δυνατό. Εγώ δεν έχω καμιά περίπτωση υπόψη μου που το να πάρει το ποδήλατο κανείς μαζί δυσχεραίνει τον άνθρωπο, δυσχεραίνει το ταξίδι με συγχωρείτε πολύ. Μπορεί να συμβαίνει αυτό για μεγάλες ομάδες που έχουν να πάρουν πάρα πολλά ποδήλατα μαζί. Υπάρχει όμως στη Γερμανία ο ICE4, το, το σιδηρόδρομος αυτός, ο οποίος επιτρέπει ε, να παίρνουν μαζί τα ποδήλατα. Και μάλιστα έγιναν και ειδικέ προμήθειε εξοπλισμού για να ε, μπορέσει να ανταποκριθεί στι ανάγκες αυτές. Και αυτό έχει νόημα για το σιδηρόδρομο, διότι και στο αεροπλάνο μπορώ να πάρω το ποδήλατό μου μαζί και σε ορισμένες ε, λεωφοριακές γραμμές. Στα λεωφορεία έφτασαν τα τελευταία χρόνια από 15.000 ποδήλατα το χρόνο σε πάνω από 100.000. Γνωρίζουμε ότι τα τρένα δεν είναι γεμάτα. Όσα λοιπόν λένε ως τώρα σειρόδρομοι για να αποφύγουν, για να αποφύγουν την υποχρέωση αυτή είναι εντελώς παράλογα. Ε, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ανέβει σε ποδήλατο ποτέ τους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση που βεβαίω και έχει βελτιώσει το κείμενο τη Κομισιόν το σημείο αυτό, θα συνεργαστούμε ευχαρίστως μαζί σα και για μα προτεραιότητα έχει ο επιβάτης και όχι η σιδηροδρομική επιχείρηση. Και μια τελευταία φράση, όταν ο κ. Γκρούμπε παρετήθηκε από το σιδηρόδρομο, ε, το λέει σήμερα η εφημερίδα, έλαβε 2,3 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση επειδή δεν βρίσκεται πλέον στη δουλειά του με 2,3 εκατομμύρια θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν για 10 και 15 χρόνια την ανωτέρα βία. Αυτά ήθελα μόνο να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιλόνεν θέλει να λάβει το λόγο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και, και εσείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θερμές ευχαριστίες στον Μπόγκουσλαβ Λιμπεράτσκι για το για την ε, έκθεσή του. Το πιο σημαντικό είναι να βάλουμε όντω τον επιβάτη πρώτο. Έτσι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους επιβάτες στον σιδηρόδρομο. Να χρησιμοποιήσουν δηλαδή περισσότερο οι άνθρωποι τον σιδηρόδρομο. Υπάρχουν μερικά πράγματα στην εκθεσή του που είναι σημαντικά για μας, όπως η προσβασιμότητα, η ασφάλεια, η ευελιξία από την πλευρά του επιβάτη. Όταν θα έχουμε ένα ανοιχτό διαφανές σύστημα όπου ο επιβάτης πραγματικά είναι η προτεραιότητα, τότε μπορούμε να οργανώσουμε πραγματικά σωστά τις υδρομικές υπηρεσίες που πραγματικά θα έπρεπε ήδη να τις είχαμε σε όλη την Ευρώπη σήμερα. Ας συνεχίσουμε την συνεργασία και είμαι βεβαία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές λύσεις. Νομίζω ότι με συνεργασία θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις που να εξυπηρετούν τον στόχο. Ευχαριστώ κυρία Κιλόνιν και βεβαίως ε, σημειώνω την αισιόδοξη στάση σας. Θα αναγκαστώ να περιορίσω λίγο τον χρόνο σας από εδώ και εμπρό γιατί έχουμε κάποια καθυστέρηση. Κύριε Μπάρ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πρότασή του. Ήδη την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε και είπα ήδη στον Μπόγκουσλαβ, ο οποίος προσπαθεί να έχει μια ισορροπημένη προσέγγιση, θεωρώ όμως θα μπορούσε να είχε φανεί πιο θαραλέος η ενημέρωση και η φροντίδα για τον επιβάτη έρχονται πρώτα και ιδίω στην αλυσίδα του ταξιδιού που αποτελείται δηλαδή από διάφορα τμήματα πρέπει εκεί να είναι ασφαλής σε όλη τη διάρκεια ο επιβάτης. Άλλο θέμα είναι η συμπερίληψη του, των διαμεθοριακών αλλά και των διεθνών μεταφορών που εκεί θα πρέπει να αποφύγουμε να προκαλέσουμε περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια. Δηλαδή να κατασκευαστεί το ολόκληρη, ε, να γίνει ολόκληρη κατασκευή μόνο για να πάρει λίγα ευρώ εν τέλει ο επιβάτης νομίζω δεν αξίζει τον κόπο. Θα πρέπει να μπορούν οι επιβάτες να αγοράζουν το εισιτήριο βέβαια και πάνω στο σειρμό και για, τα, για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες ή με δυσκολίες στην κινητικότητα Εκεί πρέπει, συμφωνώ και εγώ, να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος προειδοποίησης. Για περιπτώσεις ανωτέρας βίας αυτό δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε μείωση του επίπεδου προστασίας του καταναλωτού. Συμφωνώ επίσης με την προσπάθεια εναρμόνισης και με άλλες, άλλους κανόνες των μεταφορών και θα κάνω και σχετικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό και τριάντα δεύτερα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να τηρείτε τον χρόνο σας. 1 και 30, κυρία Άντερσον. Δεν έχει μικρόφωνο η πρόεδρος. Κύριε Άντερσον, εσείς. Από ό,τι κυρία Ροβουνταλόν. για την εφαρμογή του, τέρτου, του τέταρτου πακέτου ε, των σιδηροδρόμων. Αναμένεται η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους συμπολίτε μας. Έχουμε δηλαδή την ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται μόνο με, την, με το ξύλωμα των κρατικών μονοπωλίων, αλλά και με την προστασία των επιβατών. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Η έκθεση που μας υποβάλλει θα πρέπει να ενισχύσει τις φιλοδοξίες μας για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Δεν είναι αποδεκτό ο κανονισμός να μην λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές συνδέσεις που γίνονται ε, με, σε συνεργασία με το δημόσιο. Ενώ τώρα, μέχρι τώρα αποκλείονται και αποτελούν μεγάλο αριθμό των επιβατών. Είναι οι καθημερινοί επιβάτες, οι οποίοι κινούνται δηλαδή σε κοντινές αποστάσεις και ε, για να πάνε στους δουλειές τους. Θα καταθέσω λοιπόν τροπολογίες για να περιληφθούν αυτές οι συνδρομικές συνδέσεις στην ρύθμιση και να μπορέσουμε να δείξουμε στους συμπολίτε μας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μεγάλων σιδηροδρομικών εταιριών, αλλά τα δικαιώματα των επιβατών. Σας ευχαριστώ κύριε Αρεβό Νταλόν. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα ανταγωνιστικό λοιπόν. Ίσως είναι λοιπόν σωστό τον επιβάτη από χρήστη να τον κάνουμε καταναλωτή, πελάτη απαλαία συζήτηση μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και ιδιωτικών υπηρεσιών. Θα μπορέσουμε να δώσουμε όχι δικαιώματα, αλλά να τους επιτρέψουμε να ασκήσουν την εξουσία τους οι επιβάτες καταναλωτές. διότι εν τέλει η τιμή του, το αντίτιμο του εισιτηρίου συμβάλλει εν μέρη μόνο στη λειτουργία του συστήματος. Τώρα, δύο πρακτικές παρατηρήσεις. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να επιτρέψει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός επιβατών που θα επιτρέπει να συλλέγονται οι αποζημιώσεις, τα νέα εισιτήρια και να αποφευθεί βέβαια να καταφέρουν στα δικαστήρια για ποσά της τάξης των 25, των 8 ή των 2 ευρώ όταν υπάρχει καθυστέρηση 30 λεπτών για ένα εισιτήριο το οποίο κοστίζει 50 ευρώ. για τις ε, μεταφορές θα μπορέσει να τους δοθεί ένα εμπορικό καθεστώς όπως και στις αεροπορικές εταιρείες. Θα πρέπει να απαγορευτεί όπως συμβαίνει τώρα οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να θεωρούν ότι τα ε, τιμολόγια τους και τα οράλια τους είναι επαγγελματικό μυστικό και ότι εν τέλει ο ανταγωνισμός βασίζεται στη δυνατότητα σύγκρισης. Χρειάζεται ένα ανοιχτό σύστημα όπου οι εταιρείε θα αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό και τέλος, μιας και μας δίνεται λίγο χρόνο, μιλούμε, μιλούμε πολύ για τις ελλείψεις και για τις ελλείψεις αισθήσεων. Αν είναι κάποιος τυφλός για παράδειγμα, άντε τώρα να βρείτε τα κλειδιά για να μπείτε στο αυτοκίνητο και μέσα στο όχημα να μπορέσετε να βρείτε τη θέση σας. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ. Δεν αφισβητούμε την προσήλωση του εισηγητή στον τομέα το σιδηροδρομικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο και από αυτήν άποψη ενδιαφέρουσα έκθεση. Να πω όμω με κάθε σεβασμό ότι μπορούμε και καλύτερα και συμφωνώ με τα σχόλια του κύριου Βανίλ Τσέμπα και του κύριου Μουζελιέ και άλλων. Γιατί νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να βάλουμε τον επιβάτη στο επίκεντρο του ζητήματος και το απαιτούν αυτό από εμά οι ευρωπαϊκές συνθήκες όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Να ρωτήσω λοιπόν τον εισηγητή τι είχε κατά νου, ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό, γιατί μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικαιωμάτων των ε, Επιβατών μια επιστολή που αναφέρει ακριβώς ότι απορρίπτουν την πλειοψηφία των τροπολογιών του εισηγητή. Θα του ζητούσα λοιπόν να το ξανασκεφτεί σε περίπτωση ας πούμε ανωτέρας βίας. Ε, νομικά αυτό που προσπαθεί να κάνει αντιστρέφει ε, και ακυρώνει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό να κάνει η Επιτροπή μας, γιατί νομίζω ότι η λύση του δεν επιτρέπει μια ενδιάμεση λύση, κάτι το οποίο επιτρέπει η Κομισιόν. Και ο κύριος Μουζιβιέρ θεωρώ ότι έχει κάνει σωστά σχόλια εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε εδώ μια ενδιάμεση λύση και να δούμε τι γίνεται με, την, με τις προειδοποιήσεις όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα εστήρια ας πούμε, σε μεγάλους σταθμούς, ίσως κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι γίνεται καλή την πίστη αυτό, αλλά εκπλήσωμαι και απογοητεύομαι και διαδικαστικά Πρόεδρε, να πω ότι εδώ έχουμε κάτι το νέο, ιδιαίτερα μετά από τα νέα σχολεία και μετά από την έλλειψη χρόνου. Μήπως θα μπορούσαμε να πάμε πάλι στην ΙΜΚΟ και να δούμε τι γίνεται με το Προεδρείο της, να το θέσουμε εκεί επιγόντως, ώστε να θεωρηθούν οι καταναλωτές εδώ επιβάτες, οι επιβάτες καταναλωτές και σε αυτήν την περίπτωση ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Άντερσεν. Υπενθυμίζω ότι μένουν ακόμα τρει εβδομάδε διαπραγματεύσεων και συμβασμών. Έχουμε ακόμα χρόνο λοιπόν για συζήτηση. Κύριε Τελίσκα, έχετε, θέλετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω το μήνυμα που έστειλαν και άλλοι, γιατί βλέπω και συνάδελφοι και από άλλες πολιτικέ ομάδε, σοσιαλιστές και αλλού, στέλνουν το εξή μήνυμα, ότι πολλά από αυτά που αναφέρει η έκθεση ανατρέπουν Δεν πρέπει μόνο λοιπόν να χάσουμε εδώ ευκαιρίε. Θα ήθελα λοιπόν ο συνάδελφο να επανέλθει, ο συγητή, να επανέλθει με μια πιο φιλόδοξη έκθεση, ώστε να βάλουμε στο επίκεντρο πραγματικά του επιβάτε ω καταναλωτέ ώστε να έχουμε περισσότερα στο μέλλον, όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα, αλλά και στον ε, πολυτροπικό τομέα των μεταφορών. Εδώ ας πούμε, μιλάμε μάλιστα και για ένα τρόπο μεταφορών, τις δρομικές μεταφορές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος, ο κύριος Τενίσκα. Πίζαν Κολόν, καλημέρα. Κύριε Κολόν, για πείτε μας την άποψη της ε, ΟΚΕ okay, για τρία λεπτάκια. Σας φτάνει. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εργανομένη κοινωνία των πολιτών που εκπροσωπείται στην ΟΚΕ είναι πολύ ευαίσθητη για αυτό το θέμα. Έχει μεγάλη ευαισθησία γιατί σήμερα δεν γίνεται να μιλάμε για ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης αν ταυτόχρονα δεν, δεν υπάρχουν ως προϋπόθεση όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη κυκλοφορία. Οπότε εδώ χρειάζεται να κάνουμε κάποια βελτίωση. Τα στοιχεία του συγητή αποτελούν μια πηγή βελτίωσης, αλλά ίσως θα έπρεπε να πάμε παραπέρα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές τις μεγάλες εξαιρέσεις και όλες αυτές τις διατάξεις οι οποίες μου θυμιζουν καποια κάποιο opt-out που έχουν απορρίψει κατά κόρον οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οπότε θα έπρεπε για αυτό το θέμα να πάμε προς τα πάνω, προς τα ανάντι και να πάμε προς τις ε, χώρες, τις κοινωνίες, τις περιφέρειες όπου ήδη υπάρχει αρμονική λειτουργία του σιδηροδρόμου, όπου υπάρχουν διατάξεις υπέρ των πολιτών σε δύσκολες περιπτώσεις. Υπενθυμίζω αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως για την αναπηρία. Η αναπηρία που δεν είναι μόνο κινητική, αναπηρία πολλών ειδών που θα πρέπει να λεφθεί υπόψη. Και μια και είμαστε στην ψηφιακή εποχή, Πρόεδρε, μου φαίνεται παράξενο για να μην πω ότι είναι σοκαριστικό να μην μπορούμε να δώσουμε μια λύση γρήγορα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να αποζημιώνουμε, πολύ σύντομα θα πρέπει να δίνουμε εναλλακτικέ λύσει όσον αφορά στις μετακινήσεις. Τέλος, θα ήθελα να σας ζητήσω, Πρόεδρε, από όλη την Επιτροπή σα, να τηρήσουμε τις προθεσμίες, να μην αφήσουμε περάσει χρόνος γιατί εδώ έχουμε ένα μείζον στοιχείο όσον αφορά την αντίληψη της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στους πολίτες της, ιδιαίτερα αυτούς που μετακινούνται, έχετε την ευκαιρία να το κάνετε, έχετε την υποστήριξη της οργανωμένης κοινωνίας ε, των πολιτών, προχωρήστε, Είμαστε μαζί σας, σας στηρίζουμε και είμαστε πάντοτε έτοιμοι να το διατυμπανίσουμε αυτό, γιατί αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτό θα πρέπει να κάνουμε ως εκπρόσωποι. Τι αποφασιστικότητα που έχετε κύριε Κολόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΟΚΕ για την στήριξη. Ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο σας. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ελίζαμπετ Κοτός, καλωσορίσατε. Επικεφαλής της ε, Γενικής Δευθυσμού. Ε, τρία λεπτάκια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που δώσατε προτεραιότητα σε αυτό το φάκελο εδώ στην Επιτροπή σας και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Πράγματι, προσπαθήσαμε να συνδέσουμε να συνδυάσουμε όλα τα, τα συμφέροντα και των επιβατών και των παρόχων των υπηρεσιών αυτών. Αλλά θα πρέπει να πω ότι για τις επιχειρήσεις, για τις εταιρείε τις συνδρομικές, εμείς θα θέλαμε οι επιχειρήσεις αυτές, οι εταιρείε αυτές οι συνδρομικές να βοηθηθούν. Οπότε αυτό που προτείναμε, παραδείγματος χάρη, είναι το να αντιμετωπίζουν λιγότερα βάρη, ας πούμε, να υπάρχουν υπεύθυνοι υποδομών, ε, εκδοτηρίων και τα λοιπά, σταθμάρχες που θα ε, μοιράζουν αυτό το βάρος ώστε η νομοθεσία μας να μην επιβαρύνει τους ε, επιβάτες. Και πιστεύουμε ότι οι κανόνες που αφορούν το πακέτο για το σιδηρόδρομο σε κάποιε περιπτώσει είναι ελληπή. Οπότε χρειάζεται, α πούμε, ένα συντονισμό για περιπτώσει εκτακτού ανάγκη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Και αυτό είναι βεβαίω απόλυτα απαραίτητο σε περίπτωση που έχουμε σοβαρέ ε, διαταραχέ στην παροχή τη υπηρεσία αυτή. Επίση, θέλουμε να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδιαίτερα στον κανονισμό που υποβάλαμε σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση που προκάλεσε κάποιες συζητήσεις. Κατά νου είχαμε να προτείνουμε τα ίδια που ισχύουν στις αερομεταφορές, δηλαδή ότι εκπαιδεύουμε όχι μόνο τα άτομα τα οποία σχετίζονται με αυτούς που έχουν μειωμένη κινητικότητα, αλλά και αυτούς που μπαίνουν στην υπηρεσία την αντίστοιχη του σιδηροδρόμου. Γιατί αλλά λάβουμε τα υπόψη μας με αναπηρία, με μειωμένη κινητικότητα και τα, προβλήματα, τα προβλήματά τους, τότε εδώ μιλάμε για ένα συνολικό πακέτο που έχει να κάνει με τον σχεδιασμό των δωματίων, με τον καθαρισμό, με πολλές άλλες πτυχές σημαντικές και γι' αυτό ακριβώς το βάλαμε εδώ. βία τώρα. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι οι κανόνες εδώ δεν ισχύουν τους έπι, γιατί μιλάμε για ζημιά και αποζημίωση. Οπότε θεωρούμε ότι αυτοί οι κανόνες εδώ δεν ισχύουν. Και δεν θέλουμε να υπάρχει ευρεία και εκτεταμένη νομολογία που θα καθορίζει ακριβώ τι είναι συνθήκη και τι όχι. Και γι' αυτό ακριβώ θέλαμε να έχουμε ξεκάθαρες και περιορισμένες παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις που θα αφορούν κυρίως θεομηνίες και όχι ανθρώπινη παρέμβαση. Τα πλαίσια δηλαδή του ορισμού των εκτάκτων περιστάσεων. Περίπου όπως κάνουμε ακριβώς και εσάς μεταφορές στις θαλάσσιες κτλ. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχεία εδώ όσον αφορά την ευκολία εφαρμογής σε αυτό το πεδίο των μεταφορών. Και σε σχέση με τα άλλα ζητήματα που αναφέρονται, ιδιαίτερα για το ενιαίο εισιτήριο, το through ticketing, πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι λαμβάνει ο επιβάτης. Εμείς θέλουμε ο επιβάτης να είναι σε θέση να αποφασίσει τεκμηριωμένα Δηλαδή η απόφαση από το τέταρτο πακέτο για το ενιαίο ειστήριο πρέπει να προϋποθέτει μία πρώτη γνώση εκ μέρους του επιβάτη να ξέρει ακριβώ τι να περιμένει. Και αυτοί που πολλούν τα ειστήρια, οι επιχειρήσει αυτέ, οι εταιρείε αυτέ, θα πρέπει να εξηγούν ακριβώ περί τίνο εισιτηρίου πρόκειται. Γιατί πράγματι οι επιβάτε κυρίω θέλουν να μετακινούνται και να συνδέονται και όχι να περιφέρονται από εταιρεία σε εταιρεία. Γι' αυτό ακριβώ το νέο εισιτήριο είναι ένα βασικό κομμάτι εδώ όσον αφορά το κανόνα του αποτεκτικού στοιχείου σε αυτό το πλαίσιο. Και θεωρούμε ότι αυτός ο κανόνας του αποτεκτικού στοιχείου μπορεί να βοηθήσει τους ε, επιβάτες σε περίπτωση ασάφειας όσον αφορά την νομοθεσία σε σχέση με τα νέα εισιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ευχαριστώ κυρία Κοκάς για αυτά που είπατε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Λιμπεράτσκι για δύο λεπτάκια. σε σχέση με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και η ΟΚΕ και η Κομισιόν. Κύριε Λιμπεράτσικη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γρήγορα γιατί δεν γίνεται να σχολιάσω τα πάντα. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι συμφωνούν για το ότι έχουμε να κάνουμε με ένα, μια, μια πολύ σημαντική έκθεση που αφορά εκατομμύρια πιβάτες, εκατομμύρια άτομα. Μετά καταγράφω την βούληση όλων για συνεργασία και σας ευχαριστώ. Επίσης, Νομίζω ότι όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Και όπως είπε μια συνάδελφος, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους επιβάτες ως ε, πελάτες, ως καταναλωτές. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών. Η Κριστίνα Ρεβό παρουσίασε κάποιες απόψει που εκφράζουν τους σοσιαλιστές. Οπότε θεωρώ ότι αυτέ είναι δικέ του. Και τέλος, ευχαριστώ για τα καλά σα σχόλια και τα καλά λόγια. Έχω πρόθεση να προχωρήσω, έχοντας κατά νου ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τους υδρόδρομους, να έχουμε περισσότερους, περισσότερους επιβάτες και να είμαστε συνεπείς όσον αφορά την ευρωπαϊκή κλίμακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπεράζη και Λιακή πρόεδρος. Να πω και εγώ τα δικά μου. Τρίτη 27 Μαρτίου στις 11 είναι η προθεσμία την κατάθεση των τροπολογιών. Να το ξαναπώ για να το σημειώσετε. Το γράψατε, ωραία. Ωραία, προχωράμε. Λέει πρόεδρος. Με την ε, παρουσίαση από την Επιτροπή της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΔΣΕ. δηλαδή η επένδυση σε υποδομές μεταφορών βιώσιμων στην Ευρώπη είναι ένα θέμα το οποίο μας είναι προσφυλές ως Επιτροπή Μεταφορών. Μπορούμε λοιπόν τώρα να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα τα μέχρι τώρα. Κύριε Ρανόμες αφήστε τα πηγαδάκια. Αν θέλετε, μπορείτε να βγείτε έξω. Είναι λοιπόν σημαντικό για μας να μάθουμε ποια είναι τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα, να τα συζητήσουμε και να συνάξουμε συμπεράσματα σε σχέση με την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης όσον αφορά το ΔΣΕ που ξέρουμε ότι θα είναι καθοριστικό όσον αφορά τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των εργασιών. Έχουμε τον κύριο Ολιβιέ Σιά. Γεια σας. Από την Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ και πάλι της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα δώσουμε το λόγο για να κάνετε την παρουσίασή σας. Θα ακούσουμε προσεκτικά την εισήγησή σας και μετά θα κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας. Έχετε δέκα λεπτάκια για αυτή την παρουσίαση. Κύριε Σία, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό συνδέτα στην Ευρώπη που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικές εβδομάδες. Στόχος είναι να κάνουμε τον απολογισμό της πρώτης φάσης υλοποίησης του προγράμματος τα πρώτα 3,5 χρόνια και βεβαίως να δηλώσουμε διδάγματα και για την επόμενη περίοδο. Η έκθεση καλύπτει τρει ε, τομεί, μεταφορές, ενέργεια, ψηφιακά, αλλά εγώ σήμερα βέβαια θα σταθώ στο σκέλος ε, των μεταφορών. Θα ξεκινήσουμε με ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. Πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά στην υλοποίηση του προγράμματος να σας αναφέρω μόνο ένα στοιχείο στην τέταρτη στήλη. 95% λοιπόν αναφέρεται του προπολογισμού έχει ήδη κατανεμηθεί σε επιχορηγήσεις. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι το 95% του προπολογισμού έχει ήδη κατανεμηθεί μετά από 3,5-4 χρόνια υλοποίησης. Και αυτό βέβαια μεταφράζεται και σε αναλήψεις ε, πιστώσεων και πληρωμών. Σε επίπεδο λοιπόν ε, αναλήψεων είμαστε στο 40% και πληρωμών στο 60%, 16% συγγνώμη. Ιδίως αυτό το στοιχείο του 40% το επισημαίνω γιατί δείχνει ότι έχουμε έναν τρόπο διαχείρισης του προπολογισμού που μας επιτρέπει να ε, κάνουμε αναλήψεις υποχρεώσεων μόνο κάθε χρόνο βάσει της πραγματικής προόδου των επιμέρους δράσεων. Αυτό μας επιτρέπει να ιεραρχούμε εκ νέου προτεραιότητες και να διοχετεύουμε κονδύλια ανάλογα με την πρόοδο. Θα επανέλθω σε αυτό στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατανομή, όπως ξέρετε, ο κανονισμός F καλύπτει Ευρέωσε τον τομέα των υποδομών, αλλά προσδιορίζει και συγκεκριμένες προτεραιότητες που βεβαίως έχουμε τηρήσει. Βλέπετε ότι στις η διασυνεριακή διάσταση του προγράμματος είναι εξαιρετικά σημαντική. 66% του συνολικού προπολογισμού πήγε στους ε, διαδρόμους, ε, τους βασικούς διαδρόμους, Core Network Corridors, και σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά συστήματα όπως το ETMS πήρε πάνω από ένα δις περίπου, το CESAR 1,3 δις. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μεγάλο τμήμα ε, του προπολογισμού, η μερίδα του λέοντος, πηγαίνει σε αυτή την πανευρωπαϊκή διάσταση των δικτύων. Να τονίσω επίσης ότι μεταξύ των διαφόρων ε, προτεραιοτήτων έχουμε και την καινοτομία που έχει αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο πλέον τα τελευταία χρόνια. Από τότε που ξεκινήσαμε ειδική έκκληση και για τα εναλλακτικά καύσιμα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο του προβλησμού που μάλλον θα αυξηθεί. έχουμε οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία, μια νέα κατανομή του υπερπολογισμού για να λάβουμε υπόψη ε, την εξέλιξη των ε, προτεραιοτήτων πολιτικής και βέβαια την ε, απεξάρτηση από τον άνθρακα και η ψηφιοποίηση. Εδώ είναι δύο σημαντικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ανά τρόπο μεταφοράς. Και πάλι δεν προκαλεί έκπληξη ε, το γεγονό ότι κατά συνέπεια των κανόνων επιλεξιμότητα του ΣΕΦ, το μεγάλο τμήμα του προπολογισμού πήγε στι ε, σιδεδρομικέ υποδομέ και στις, ε, στην εσωτερική νευσεπλοεία. Τα οδικά δίκτυα και οι αεροπορικές μεταφορές ε, συνδέονται αυστηρά με, τη, με τα ψηφιακά στοιχεία ή με στοιχεία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αυτών των ε, των τρόπων μεταφοράς. Το ίδιο ισχύει και με την ναυτιλία και με την πολυτροπική, τις πολυτροπικές μεταφορές. Επομένως, ε, κατά κύριο λόγο, βασιζόμαστε σε ε, βιώσιμες, βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Σε ό,τι αφορά τώρα την συμπληρωματικότητα με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, να επισημάνω το αδερφάκι του ΣΕΦ, το ERDF και το Ταμείο Συνοχής. Αυτά τα δύο προγράμματα είναι τα αδερφάκια λοιπόν ε, ε, του ΣΕΦ, τα πλέον ε, συγγενή προγράμματα. Αν δείτε τη στήριξη προς το βασικό δίκτυο, συνολικά έχουμε 40 δις καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος. 23 προκύπτουν από το ΣΕΦ, τα υπόλοιπα από το Ταμείο Συνοχή 13 και από το ERDF έχουμε 4 δις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό δεν δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα αλληλεπικαλύψεων ή έλλειψη συμπληρωματικότητα. γιατί το ΣΕΦ βασίζεται σε διασυνοριακά στοιχεία και στο σιδηρόδρομο κατά βάση, ενώ το Ταμείο συνεχίσει και το ERDF καλύπτουν και άλλα ε, τμήματα του, των δικτύων. Όμω, ιδίω για το σιδηρόδρομο υπάρχει μερική αλληλεπικάλυψη, την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η συμπληρωματικότητα προς το πρώτο διασφαλίζεται στο αρχικό προγραμματικό στάδιο και κατά τη διάρκεια επιλογής όπου συνεργαζόμαστε με συναδέλφου από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών και σε κάποιο βαθμό σε ό,τι αφορά και την ε, σύγκληση των κανόνων. Αυτό είναι το σημείο που έχουμε επισημάνει στην αξιολόγηση ως ε, θέμα που επιδέχεται βελτίωση. Για το χρηματοδοτικό μηχανισμό και τη συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, πρώτα είχαμε το ΣΕΦ και μετά το ΕΦΣΥ από πλευράς χρονικής αλληλουχίας. Και γι' αυτό πολλά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί υπό το ΣΕΦ στη συνέχεια προχώρησαν ε, μέσω του ΕΦΣΥ. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε να συγχωνεύσουμε επιμέρ, ε, τα επιμέρους ε, χρηματοδοτικά εργαλεία σε ένα ταμείο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σίγουρα η κατεύθυνση που πήραμε από το ΣΕΦ με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία Προ το ΕΦΣΙ και προς άλλα μεγάλα ταμεία, αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά τις ε, μορφές ε, χρηματοδότηση. το ΣΕΦ χρησιμοποιεί επιχορηγήσει κατά βάση. Έχουμε εδώ το γενικό συνολικό φάκελο και τον φάκελο συνοχής των 11 εκατομμυρίων. 11 δισεκατομμυρίων μάλλον, έχουμε την ε, μέγιστη και την βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων μέσω της αρχής use it or lose it. Δηλαδή είτε αξιοποιεί κανείς τα κονδύλια είτε τα χάνει. Δεν ε, δεσμεύουμε το σύνολο ε, του ποσού από την αρχή του προγράμματος και έτσι είμαστε στη δυνατότητα να διορθώσουμε, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη με, μέσω της τροποποίησης ε, της συμφωνίας επιχορήγησης. Και έτσι μπορούμε να δεχθούμε σε μείωση του ποσού, αν δούμε ότι ε, δεν υπάρχει σωστή απορρόφηση. Και αυτό μας επιτρέπει, αν το κάνουμε αυτό εγκαίρως, να επαναδιοχετεύσουμε τα κονδύλια σε άλλα προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτή η αρχή ε, δεν λειτουργεί τιμωρητικά μιλούμε για χρήματα που έτσι και δεν πρόκειται να απορροφηθούν από αυτό το πρόγραμμα. Οπότε είτε θα χαθούν τελείω, είτε έχουμε δυνατότητα να τα επαναδιοχετεύσουμε αλλού, ε, να στηρίξουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Χρησιμοποιούμε και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Ήδη ανέφερα ότι το ΣΕΦ ήταν ε, ένας πρόδρομος αυτού του συστήματος και οδήγησε στην ε, δημιουργία του ΕΦΣΙ από το 2015 και ε, πειραματιζόμαστε και με τη χρήση του blending, δηλαδή χρησιμοποιούμε επιχορηγήσεις σε συνδυασμό με άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και σας ε, δείχναμε τα αποτελέσματα του πρώτου εγχειρήματο το Δεκέμβριο με ευρύτερη συμμετοχή πολλών ε, ε, εθνικών τραπεζών, ακόμα και εμπορικών, με σκοπό την συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, ε, σίγουρα δεν μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα, γιατί από πίσω έχουμε βέβαια την πολιτική τεντή. Χρειαζόμαστε λοιπόν ξεκάθαρο προγραμματισμό στο πλαίσιο TNT, στο πλαίσιο των διαδρόμων, συντονισμός και όλο αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευρύ ε, πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αναλάβει στη συνέχεια το ΣΕΦ. Έχουμε την ε, διαδικασία επιλογής. Έχουμε πολύ περισσότερα προγράμματα που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πλέον και αυτό είναι θετικό. Γιατί έτσι επιτρέπουμε την επιλογή των πλέον ανταγωνιστικών προγραμμάτων, των πλέον όριμων προγραμμάτων που έχουν και προσταθεμένη αξία. Αυτό είναι και το κέριο μήνυμά μου, συμπερασματικά, ότι το ΣΕΦ είναι ένας μηχανισμός που συνάδει πλήρως με τους στόχους πολιτικής μας ό,τι αφορά την διασύνδεση, την αυξάτηση από τον άνθρακα και την ψηφιοποίηση. Έχει προσθεμένη αξία γιατί για τα προγράμματα που δεν θα λάμβαναν χρηματοδότηση είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε, με όρους αγοράς, λαμβάνουν στήριξη από το ΣΕΦ και Βέβαια μιλούμε για δημόσια αγαθά ευρωπαϊκών διαστάσεων. Κλείνοντας, ε, να υπενθυμίσω ότι ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο της υλοποίησης. Έχουμε δύο εκκλήσεις που τρέχουν προς το παρόν, δύο διαγωνισμούς, ένα για το ΣΕΖΑΡ στον ε, τομέα της αεροπορίας μέχρι τον Απρίλιο τρέχει και η δεύτερη φάση του blending επίσης κλείνει τον Απρίλιο με σημείο εστίαση στα εναλλακτικά καύσιμα. Ε, τέλος, ε, προετοιμάζεται ακόμα ε, ένας διαγωνισμός για τα εναπομείναντα κονδύλια με επίκεντρο ε, την διασύνδεση και την πολυτροπικότητα στο πλαίσιο του, της τρίτης δέσμης κινητικότητας. Όλα αυτά τα στοιχεία και σε ό,τι αφορά και το μέλλον ε, της διαδικασίας θα βρεθούν στο επίκεντρο του επόμενου δεκαήμερου στην εκδήλωση που θα λάβει η χώρα στη Λιουμπλιάνα στα τέλη Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος, για την παρουσίαση. Απευθείας θα περάσουμε στη συζήτηση. Δύο λεπτά θα έχετε στη διάθεσή σας ο κύριος Βιμ Κάμπ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετικά ξεκάθαρη αυτή η παρουσίαση. Ελπίζω να έχει ήδη κλείσει το δωμάτιο ο εκπρόσωπος της Επιτροπής από, στη Λιουμπλιάνα. Εγώ το έκανα πάντως. Θα ήθελα να λάβω και γραπτό αυτή την παρουσίαση, γιατί είμαι παλαιάς κοπής και μου αρέσει να τα βλέπω μπροστά μου τα στοιχεία. Και η κυρία Αιάλα Ζάντερ, με την οποία συχνά συμφωνώ, με στηρίζει σε αυτό το αίτημά μου. Τώρα περάσω στα πιο δύσκολα. Τι δεν κατάλαβα. Τι είναι ο πολλαπλασιαστής του ΣΕΦ ποιος είναι έχουμε την επιχορήγηση, αλλά μετά φαντάζομαι πρέπει να υπάρχει και ένας πολλαπλασιαστής ε, με εθνική συνεισφορά, blending, εύση. Ενδεχομένως παρουσιάζεται τα στοιχεία, λέτε 27 δις έχουμε δώσει, αλλά ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής. Δεύτερον, λέτε use it or lose it. Η αρχή που αναφέρατε αυτό συνδέεται με κάποιο, κάποια χρονική προθεσμία. Γιατί μας παρουσιάσατε την αρχή, αλλά υπάρχει κάποιο όριο οπότε επιστρέφονται τα κονδύλια εάν δεν απορροφηθούν. Και μετά πηγαίνουν και πάλι σε call, πάλι σε διαγωνισμό, δηλαδή τα κονδύλια. Πότε ακριβώς ε, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του use it or lose it. Και δεύτερον, ποια είναι η διαδικασία επαναδιοχέτευσης των κονδυλίων. Μετά, δεν άκουσα τίποτα για την αστική διάσταση. Έχει γίνει κάτι στην πόλη ή όχι. Ή δεν μπορείτε να το πείτε. Δεν μπορείτε να κρίνετε. Γιατί αυτό το urban, η αστική διάσταση, είναι η νέα πρόκληση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εύση τώρα. Κάθε φορά μιλούμε θετικά για το εύση. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας πει τι έχουμε πετύχει τελικά με το εύση. Για παράδειγμα, σε σχέση με το πρώτο μου ερώτημα, ποιο είναι ο πολλαπλασιαστής του ΣΕΦ. Γιατί όλοι λένε τα καλύτερα για το ΕΦΣΙ, αλλά ποτέ δεν έχουμε δει τι συμβαίνει στην πράξη. Τέλος, υποθέτω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει αυτή την ε, παρουσίαση ως ε, ένα εξαιρετικό κίνητρο για τις μελλοντικέ ε, διαπραγματεύσεις για το πει. Γιατί με τέτοια στοιχεία θα είναι σε καλή θέση ο κύριος Έντεγκερ. Δεν ξέρω η DG Move τι γνώμη έχει γι' αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμπ. Κύριε Ερτίκ η κυρία Γιάννα Σέντερ θα ε, αναπτύξει την θέση της ομάδας μας, κυρία Πρόεδρε. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την παρουσίαση. Καταρχάς, να πω ότι θα θέλαμε και εμείς να δούμε γραπτό στην εισήγηση της Κομισιόν, να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να πω ότι ο εκπρόσωπο τη Γενική Διευθύνση MOVE είπε ότι χαίρεται που υπάρχουν πολλά προγράμματα ώστε να επιλέξει κανεί. Νομίζω ότι εν ώψη του τη σύγκρουση τη δημοσιονομική αυτό θα πρέπει να το ξαναπούμε γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και όχι προγράμματα. Χρήματα τα οποία όχι μόνο δεν φτάνουν για τα προγράμματα αλλά μπορούν να περικοπούν. Οπότε καλύτερα να αλλάξουμε τροπάριο και να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, τουλάχιστον το λιγότερο. Μετά για τους δύο διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για τα 350 εκατομμύρια για το 2018. Στην διαμέση αξιολόγηση που ήταν ουσιώδης υπάρχει αφενός αυτή και αφετέρου τα ποσά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Με Αυτό το κοιτάτε ή όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Είχαμε να δεις τελικά που δεν χρησιμοποιήθηκε. Γιατί θα θέλαμε αυτός ο τελικός διαγωνισμός να προετοιμάζεται για τις μελλοντικέ και να καλύπτει τις μελλοντικέ προκλήσεις και τις δημοσιονομικές. Για το μέλλον τώρα. ακούσαμε για την στήριξη των κυβερνήσεων και τη δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια προγράμματα αύξησης του επίπεδου συγχρηματοδότησης της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης. Δηλαδή να πάμε πέρα του 40% ευρωπαϊκής συμβολής και συγκεκριμένα προγράμματα μεγάλης προσθέμενης ευρωπαϊκής αξίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη συζητιέται και μπορούμε να το βαθύνουμε. Να πω επίσης ότι την προηγούμενη φορά είχαμε μεταφορές ενέργεια και τηλεπικοινωνίες και αυτό το τρίδημο και το Κοινοβούλιο επέμενε στο να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των τριών τομέων γιατί ο ένας τομέας επηρεάζει τον άλλον ενέργεια, ψηφιοποίηση, νέα καύσιμα, νέες μορφές ενέργειας κλπ. Η Κομισιόν μετά την ενδιάμεση και τη δεύτερη διαλογή θεωρεί ότι θα υπάρξει ένας τέταρτος πυλώνας με συνέργειες όπου θα μπορούσαμε ας πούμε, να εντάξουμε τα νέα καύσιμα για τα νέα οχήματα. Κάτι που πέρασε στην Ολομένια μετά από πρόταση του κ. Βερτού. Και μάλιστα είχαμε προϋπολογίσει 24 δις. Έχει γίνει και προκατακτική μελέτη γι' αυτό. Δηλαδή να έχουμε ένα, ξαναλέω, πυλώνα όπου θα υπάρχουν αυτές οι συνέργειες μεταξύ μεταφορών, ενέργειας κλπ. ώστε να προχωρήσουμε. Επίσης, μπορείτε να μας δώσετε μια μελέτη για την απόδοση όλων αυτών των κονδυλίων από το ΕΦΣΥ γιατί θα θέλαμε από τα στοιχεία μας δώσατε να καταλάβουμε ποια είναι η απόδοση καθαρά των μεταφορών σε σχέση με τον ορίζοντα 2020. Κατά πόσο αυξομοιώθηκαν τα κονδύλια στα διαφορετικά ταμεία, εύση κλπ. Δηλαδή, ξαναλέω, ποια είναι η απόδοση, ποια είναι η απόδοση αυτών των κονδύλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεντέρ. Ισμαέλ. Σα έδωσα για το δικό του χρόνο. Και ο Λίσκα, ο κύριε Λίσκα, ο λόγο σε εσά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπάσω, Πρόεδρε, να είμαι σύντομο. Ο Επίτροπος συζήτησε το θέμα τα θέματα αυτά μαζί μα και νομίζω ότι συμμετείχα και εγώ και ελπίζαμε του πω ότι θα είχαμε καλή έκφαση. Πάντως υπάρχουν δύο τρόποι υποβολή μιας έκθεσης. Μια έκθεση περιγραφική με πολλά στοιχεία, αριθμού, με ωραία ποσοστά κατανομή, άνοιξη υποχρεώσεων, πιστό πληρωμών και μετά γραφήματα με τις κατανομές, τις επικαλύψεις κτλ. Ωραία αυτά, αλλά υπάρχει και καλύτερος τρόπος Δηλαδή μια σοβαρή αξιολόγηση. Να δούμε κατά πόσο η αποθρακοποίηση, η ψηφιοποίηση λοιπά, αυτή η στόχη αν ρωτήσει η Δημοσιονομική Αρχή αν θα δαπανίσω ε, αυτά τα χρήματα ε, για το μέλλον και χρειαστούν περισσότερα, τι θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε ότι υπάρχουν περισσότερα προγράμματα και χρειάζεται χρηματοδότηση. Αυτό δεν φτάνει όλοι μας και οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε καλύτερη ε, συνδεσιμότητα και να ποσοτικοποιήσουμε, ας πούμε, η απαθρακοποίηση. Τι γίνεται με τα προγράμματα που ολοκληρώνονται, χρηματοδοτούνται, αλλά ποιε είναι οι προσδοκίε. Και το ίδιο και για την ψηφιοποίηση. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα στην έκθεση. Επ' αυτού και δεν άκουσαμε και τίποτα από την παρουσίαση τη Κομισιόν. Δεύτερη παρατήρηση η διάδραση με άλλα οικονομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ποια αξιολόγηση όμως γίνεται εδώ. Κοντήλια, συνοχής, το εύση, αξιολόγηση. Τι είναι όμως με τα ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να υπάρχει υψηλή προσθέμενη αξία και συνδυασμή. ώστε να δούμε τέλος πάντων υπάρχει κάποια ιδέα του ότι μπορούμε να προσδεκάμε από αυτό δεν άκουσαμε και πάλι τίποτα σχετικά. Ωραία. Καλό να χρησιμοποιούμε αυτά τα κονδύλια. Αλλά ας πούμε για τις τηλεματικές μεταφορές. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα της χρήσης αυτών των κονδυλίων. Ανάλογα με το ποσοστό χρήσης τους. 60-70-80-100%. Το Σεζάρ. Θαυμάσιο. Αλλά και πάλι, ποια πολιτική αξιολόγηση κάνουμε του ΣΕΖΑΡ. Οπότε, Πρόεδρε, καλή έκθεση σε σχέση με τα δεδομένα του παρελθόντος, αλλά αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε και να έχουμε είναι μια έκθεση που θα παράσχει μια σοβαρή αξιολόγηση ανακριτήριο και αναστόχο που έχει θέσει η Κομισιόν, με συγκεκριμένη περιγραφή και αν γίνεται και με ποσοτικοποίηση. Αυτό λείπει και αυτό θα πρέπει να κάνει η Κομισιόν. Δηλαδή, να υποβάλει σοβαρά στοιχεία σε σχέση με το επόμενο που Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Κύριε Νταλούντε, δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σύντομα. Για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Εγώ ανησυχώ. Γιατί πολλές χώρες μπορούν να παραβλέψουν ακριβώς τις επενδύσεις στην υποδομή. Οπότε ρωτάω πώς εμείς εφαρμόζουμε τα κριτήρια ώστε να διασφαλίσουμε ότι με τα κοινωνικά χρήματα θα χρηματοδοτήσουμε υποδομές που δεν όχι μόνο που δεν χρηματοδοτούν οι χώρες μέλη, αλλά για να δημιουργήσουμε και ένα εύρωστο και ισχυρό ε, δίκτυο διασυνοριακό, το οποίο θα αφορά στις μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στρικέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να μην μιλήσω για αποτελέσματα. Δεν θα μιλήσω για τον μηχανισμό τον ίδιο, συνδέοντας την Ευρώπη, αλλά για τα αποτελέσματα. Είπε κάποια πράγματα η Κομισιόν για τα προγράμματα τα μακρόπνοα που εξεγγίσαν πριν από κάποια χρόνια. Υπάρχει δυσκολία στο να παρουσιάσουν λειτουργικά αποτελέσματα. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω εν επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Αλλά θα μιλήσω για το μηχανισμό. Και θα ήθελα να επιθυμήσω ότι το συνδέοντας στην Ευρώπη αποτελεί ένα εργαλείο χρηματικής διακυβέρνησης το οποίο περιείχε τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί συν 11 δισεκατομμύρια και τα οποία μετακινήθηκαν. Οπότε το πρόβλημα εδώ δεν είναι τα χρήματα. Γιατί από αποτελέσματα είχαμε αποτελεσματικά, μάλλον θεματικά αποτελέσματα. Εσείς είπατε ότι θα πρέπει να πάμε από το, συνδέοντα, από το στην Ευρώπη προς το ΕΦΣΥ ε, συνδέοντας την ε, Κομισιόν με αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά ειλικρινά το καταλαβαίνω αυτό γιατί το να διασφαλίσουμε την ποιότητα αυτού του μηχανισμού σημαίνει ότι θα έχουμε την ε, συμμετοχή την κεντρική της Κομισιόν με την πραγματογνωμοσύνη της, την, τεχνο, τεχνογνωσία ε, της και την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης, της συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Παιδίου στον τομέα των μεταφορών είναι απογοητευτικά. Οπότε το ΕΦΣΥ πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά και πρέπει η Κομισιόν να υπερασπιστεί ένα εργαλείο Και επιθυμίζω εδώ ότι είχαμε 26 δισεκατομμύρια ε, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς ε, τι έχουν γίνει και αποτελέσματα που δεν έχουμε δει για τις μεταφορές. Οπότε ένα πολύ ωραίο εργαλείο έχουμε με το ΕΦΣΥ. Οπότε ρωτάω ποιο είναι το μέλλον, όχι μόνο το ποσοτικό στα πλαίσια ενό ε, προπολογισμού, ο οποίο εντάξει θα έχει περικοπέ, έστω και αν είμαι αισιόδοξο, αλλά θα έχουμε μια δεύτερη εκδοχή και θα βελτιώσουμε, θα τροποποιήσουμε ή θα διατηρήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο που ήταν αποτελεσματικό ή θα κάνουμε διάφορες πονηριές ε, με μεταφορές σε ε, ε, κοντιλίου που θα, διαχειριστούν από άλλους οργανισμούς από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και με τον αντιπρόεδρο αυτό το ζήτημα, θα πρέπει ενδεχομένω να επανέλθουμε. Η σχέση για την τελεματική στι ε, μεταφορέ και το συνδέοντα στην Ευρώπη είναι το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω. Οπότε θεωρείτε ότι μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Τώρα για το μέλλον. Το θέμα δεν είναι ε, αν θα έχουμε χρήματα ή όχι, αλλά τι θα κάνουμε με αυτόν τον κανονισμό πώς μπορείτε να τον βελτιώσετε και πώς θα μπορούσατε να τον προστατεύσετε από την υποβάθμιση από, αυτούς τους ε, κανονιστικ... από αυτό το κανονιστικό χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Δεν, δεν σεβαστήκατε καθόλου το χρόνο αγορεύσεώς σας, αλλά για μια φορά σας ε, το επιτρέπω. Κύριε Δεγκράντης, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που μας ενημέρωσε. Δεόντως, σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού που είχε δημοσιευθεί στις 13 του Γενάρη. Μας είπαν λοιπόν πώς εξελίχθηκε, πώς πήγε αυτός ο μηχανισμός και κατά πόσο αυτή η αξιολόγηση θα επιτρέψει το σπάτι την ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων. Αλλά μας έρχεσαν και ένα κρύο ντουζ μετά από αυτά που είπε και η κυρία Γέλα ότι μας είπαν ότι είχαμε περισσότερα προγράμματα από την κονδύλια. Αλλά όταν αποφασίσαμε τις τους δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιήσουμε τους πάντες πολλές περιφερειές ε, προφανώς επιθυμούν την ικανοποίηση των προσοκιών τους. Και θα έχουμε και νέα αιτήματα. Και στην Ισπανία υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες, μιας και μιλάμε για διευθυνωρικά θέματα. Έχουμε τη Γαλλικία, που έχει σύνορα κοινά με την Πορτογαλία και που προσδοκά ότι τα βασικά συνδρομικά δίκτυα θα ενσωματωθούν στον Ατλαντικό διάδρομο. Και σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει να θετήσουμε μέτρα σε σχέση με, το, με την ανανέωση ή τροποποίηση ή κατάργηση αυτών των μέτρων. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια πολιτική κρίση που μου φαίνεται σημαντική σε σχέση με τις ευαισθησίες των κρατών μελών. Εδώ δεν έχουμε μόνο το κανονισμό, αλλά το 9 3 2010 που περιλαμβάνει η προβλέπεται δυνατότητα τροποποίηση των διαδρόμων. Δηλαδή ανοίγει ένα, παρά, ένα παράθυρο ευκαιριών και δυνατοτήτων, οπότε αυτή η διαδικασία θα πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πόροι, ποιε είναι οι προθεσμίε, ποια είναι τα κριτήρια για να πούμε αν ή όχι θα υπάρξουν χαμηλή πόρη και κατά πόσο οι προσδοκίες και τα αιτήματα που θα υποβληθούν θα μπορούσαν να ευοδοθούν ή απλά και μόνο εδώ αν κάνουμε εδώ πέρα φιλοσοφική συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τεγκράντης. Και έχω σημειώσει και το δικό μου όνομα στον κατάλογο των αγορητών. Μας κάνετε ε, ε Κομισιόν μια πολύ θετική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού συνδέσεων από την ποσοτική άποψη όντως βλέπουμε τα, τον αριθμό των έργων που αναμένουν χρηματοδότηση κλπ. Και έχετε δίκιο που λέτε ότι κάπου είναι επιτυχία. Αλλά ποσοτική. Αν δούμε λίγο ποιοτική, ποιοτικά τα πράγματα, εγώ παραμένω σε ιδιαίτερα κριτικό πνεύμα για τον τρόπο χρηματοδότησης και για την αδιαφάνεια απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους πολίτες. Παράδειγμα, γνωρίζετε έρχονται διάφοροι και με ρωτούν ποια είναι, ποιο είναι το σχέδιο χρηματοδότησης ε, της σύνδεσης Λιών-Τουρίνου. Και εγώ έχω πρόβλημα, διότι δεν μπορώ να τα βρω τα στοιχεία αυτά. Οι συνθήκες λοιπόν για να διεξαχθεί πραγματική συζήτηση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμα δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ασκήσει αυτοκριτική για να διαχειριστεί καλύτερα τα ε, κονδύλια στον επόμενο προγραμματισμό. Είναι σημαντικό αυτό, διότι πρόκειται για πολιτική, την οποία πάντοτε υπεστήριξε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, ήταν και στο πρόγραμμα του Ταλίν και εγώ την υπερασπίστηκα, υπερασπίστηκα τον προπολογισμό για την πολιτική αυτή με όρις μου τις δυνάμεις ενώπιον των Υπουργών Μεταφορών. Θέλω λοιπόν να προβληματιστείτε και σχετικά με την ποιότητα και όχι μόνο ε, την ποσότητα των έργων, διότι μιλούμε για την προστιθέμενη αξία, για το πώς θα διασυνδεθούν οι Ευρωπαίοι, αλλά βεβαίως από την άλλη μεριά και πώς θα, μειωθεί, ε, θα μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Είναι και αυτό τεράστιο θέμα. Ανησυχούμε από την άλλη μεριά και για τις ε, επιπτώσεις της Βρετανικής αποχώρησης και της μείωσης κινητικότητας των διαφορών δικτύων. Μιλήσατε και τι υποδομέ που πρέπει να συγχρονιστούν για την ανάγκη ψηφιοποίηση κλπ. Αλλά μπορώ να σα βεβαιώσω για ένα πράγμα. Όταν ακούμε για το πρόγραμμα ΕΦΣΙ των στρατηγικών επενδύσεων, λέμε ότι είναι και σημαντικό μέρο των χρηματοδοτήσεων που εγκρίνει η Επιτροπή Μεταφορών. Και όταν εξετάζουμε αυτό το ΕΦΣΙ σήμερα, για μας είναι σκανδαλώδε το ότι μόνο 9% των έργων αφιερώνονται στις μεταφορές. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι λοιπόν, βγάζοντας αυτά που είχα μέσα μου, είμαι βεβαία ότι θα σας δούμε στη Λουμπλιάνα, αλλά θέλω να μπορέσουμε να δράσουμε πάνω στα πλαίσια του ίδιου οράματος και να ανταποκριθούμε στα κατεπήγοντα. Καθημερινή ζωή των πολιτών, μέλλον του πλανήτη, θέματα κινητικότητας, διασυνδεμένης κινητικότητας, και τέταρτο με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πρέπει να θέσουμε επιτάπητος. Σας εύχομαι λοιπόν ε, καλό κουράγιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Σία, σας δίνω πάλι το λόγο για να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων μου. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να δώσω ορισμένα στοιχεία. Βεβαίω μέσα σε μια παρουσίαση 10 λεπτών δεν μπορεί κανείς να αναπτυχθεί σε όλο το περιεχόμενο της έκθεσης ε, αξιολόγησης. Να τονίσω ωστόσο ότι είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για αποτελέσματα μετά από δύο ή τρία έτη μόνο, διότι ορισμένα έργα άρχισαν 2014-2015, αλλά το 2016. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό ε, χρονικό χάσμα, διότι από τη μια μεριά μια αξιολόγηση στα μέσα του δρόμου δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν τα προγράμματα ή τα έργα. Δεν θα ήταν ειλικρινές ε, να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να έχουμε στη θέση μας αξιολογήσιμα αποτελέσματα όλων των έργων, για παράδειγμα για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακος. Άρα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι διαστάσεις και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τις, ε, και για την αξιολόγηση στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να έχουμε πιο στέρεους δείκτες και να μπορέσουμε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε να αξιολογήσουμε στη μέση του προγράμματος και στο τέλος του προγράμματος. Όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ασφαλώς εδώ, συνεχίζω στα αγγλικά, η αφετηρία είναι ο συντελεστής συγχρηματοδότησης. Για το γενικό φάκελο αυτός είναι από 20 έως 50% πιθανώς ο μέσος όρος να είναι κάπου μεταξύ 30 και 40%. Και για τη συνοχή είναι 85% για τις περιοχές συνοχής. Η συγχρωματότητα είναι 85%. Αυτό σας δίνει μια ιδέα για την επιρροή στις επενδύσεις. Η μόχλευση ωστόσο είναι μέρος μόνο της υπόθεσης, διότι η μόχλευση μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν εξετάσετε αν το έργο θα χρηματοδοτιόταν και διαφορετικά χωρίς την υποστήριξη αυτή το έργο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα υλοποιούνταν ποτέ ή πολύ πολύ αργότερα. Άρα η μόχλευση είναι μια, ε, ένα θέμα, αλλά η προσθετικότητα, ειδικά για τη διασύνδεση της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντικότερη από τη μόχλευση. Τώρα για το use it or lose it. Η ιδέα είναι αφής στιγμής δεν διαθέτουμε το σύνολο του ποσού που έχει ε, προβλεφθεί στην ε, σύμβαση της επιχορήγησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα, υπομένα, τα απομένοντα χρήματα και για άλλα έργα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα έργο το οποίο υποτίθεται θα ολοκληρωθεί το 2021. Θα λάβει μια παράταση διότι έχει σημειωθεί καθυστέρηση και από πάνω από την παράταση που μπορεί να λάβει γνωρίζουμε με ασφαλή τρόπο ότι ένα 20% του ποσού της αρχικής επιχορήγησης είναι πέραν του χρονικού σημείου, του ορίζοντος δηλαδή. Εάν λοιπόν δεν μπορέσουμε τι, το, τι κάνουμε, το αφήνουμε τα χρήματα στη συμφωνία, ο χρόνος περνάει, η προθεσμία περνάει και τα χρήματα επιστρέφουν στις χώρες μέλη. Με το use it or lose it τροποποιούμε έγκαιρα τη συμφωνία επιχορήγησης. Αφαιρούμε τα χρήματα που ούτως ή άλλως το έργο δεν θα μπορέσει να απορροφήσει και τα βάζουμε σε νέο πρόγραμμα εργασιών για νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να τα βάλουμε σε νέο πρόγραμμα για νέα ε, πρόσκληση ενδιαφέροντος. Για μας λέμε εκεί, απόλυτη κατακλητική ημερομηνία για να το κάνουμε αυτό θα είναι αρχές 2021. Η τελευταία δηλαδή, θα, τελευταία δηλαδή χρήσιμη πρόσκληση ενδιαφέροντος θα μπορεί να γίνει αρχές 2021. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε καθαρή εικόνα για όλες τις επαναρροές και να μπορέσουμε να κάνουμε πολλές reflow calls. Γι' αυτό ο εκτελεστικός οργανισμός μας φέτος ήδη κάνει μία σε βάθος εξέταση των χαρτοφυλακίων, όπως έγινε και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπου όλες οι δράσεις βεβαίως με στόχευση κυρίως στις μεγάλες δράσεις, εξετάζονται για να δούμε ακριβώς οι δράσεις αυτές τι μπορεί να καταναλώσουν και τι όχι στην περίοδο αυτή. Και στο τέλος του έτους ή αρχές του επόμενου έτους θα μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη ε, σειρά τροποποιήσεων για τις ε, συμφωνίες δηλαδή ε, επιχορήγησης και να βάλουμε τα απομένοντα χρήματα σε νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος που μπορεί να είναι ετήσιες, διότι αυτή η υποχρέωσή μας για το 5% για περιφερειακές διαμεθοριακές, αλλά επειδή αναμένουμε να έχουμε πολύ περισσότερες επαναρροές, reflows δηλαδή από ό,τι θα είναι αναγκαίες για αυτές τις καινούργιες προσκλήσεις, θα μπορούμε να κάνουμε και κάποιες γενικές αιτήσει για το 2019 και 2020, αναλόγως των ποσών που θα ανακτήσουμε. Αυτά είναι σημαντικά να τα έχει κανείς υπόψη του για το τέλος του 19, αρχέ. 20. Και για τις συνέργειες τώρα. Χαίρομαι που θέσατε το θέμα αυτό στη συζήτηση, διότι πράγματι πρόκειται για ένα σημείο όπου η αξιολόγηση δεν μας, δεν μας έχει δείξει καλά πράγματα, διότι δεν τα πάμε καλά εκεί, διότι η περίμετρος επιλεξιμότητας των τριών τομέων πρέπει να προσθεθεί. Αν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο το οποίο πατάει με το ένα πόδι στι στις και με το άλλο στην ενέργεια, χρειαζόμαστε επιλεξιμότητα και στους δύο τομείς. Και επομένως η επικάλυψη αυτή, είναι, το, το, το, που επικαλύπτεται δηλαδή, είναι πάρα πολύ στενό. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πραγματικέ συνέργειε και να βρισκόμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τους συναδέλφους των δύο άλλων τομέων. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική αλλαγή για την ε, της συνδέοντας στην Ευρώπη για την επόμενη περίοδο. Για το ΕΦΣΙ. Λυπούμε διότι ίσως ε, στην αρχή μου τοποθέτηση να μην μου σαφής. Η ιδέα δεν είναι καθόλου να αλλάξουμε την διαχείριση ή να πάμε από επιχορηγήσεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι επιχορηγήσεις, τα grants δηλαδή, παραμένουν και θα παραμείνουν η βασική υπόσταση της ΣΕΦ. Σήμερα έχουμε ένα, μια μικρή διάσταση χρηματοδοτικού μηχανισμού μέσα στην ΣΕΦ. Για την επόμενη περίοδο θα μπορέσουμε να την αφαιρέσουμε και να την βάλουμε στα πλαίσια ενός ενίου μηχανισμού για να αποφύγουμε ώστε να αποφύγουμε να υπάρχει πολλαπλασιασμός μικρών χρηματοδοτικών μηχανισμών κατεσπαρμένων σε διάφορα προγράμματα. Θα τα βάλουμε όλα μαζί. Αν τα βάλει κανείς όλα μαζί, επιτυγχάνει εξοικονομήσεις κλίμακος και σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική εγγύηση, το reporting, την μόχλευση και βεβαίως τους οργανισμούς που αναλαμβάνουν κατανάθεση. Δεν αλλάζουμε δηλαδή την ισορροπία, η ΣΕΦ, δηλαδή η διευκόλυνση για τη σύνδεση στην Ευρώπη, θα παραμείνει σε κράντς γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρα τη και το το, των μεταφορών. Η τοποθέτηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών θα, θα τροποποιηθεί. Και για τα ποιοτικά και τις μεγάλες υποδομές. Εδώ πρέπει να πω ότι η διευκόνηση συνδέοντας στην Ευρώπη είναι μέρος της υπόθεσης αυτής. Η υποστήριξη της Ευρώπης καλύπτει συχνά εδώ πολλές χρηματοδοτικές περιόδους και εάν για ένα μεγάλο έργο καλύπτεται, καλύπτεται εκεί και δύο και τρεις περιόδους, κανείς δεν μπορεί να αφήσει χρηματοδοτική εγγύηση για ολόκληρη την περίοδο αυτή. Για κάποια πολύ μεγάλα λοιπόν project υποδομών είναι δύσκολο να καθοριστεί εξ αρχής για πόσο θα χρειαστεί εγγύηση. Μπορούμε να βάλουμε λοιπόν το ποσοστό χρηματοδότησης για μια συγκεκριμένη περίοδο, αλλά δεν είναι εγγυημένο για την επόμενη. Προσπάθησα να καλύψω τις περισσότερες από τις ερωτήσεις και ας αρκεστώ σε αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οι απαντήσεις σας ήταν και σαφείς και πλήρης και απαντούσαν ξεκάθαρα στα ερωτήματά μας. Νομίζω ότι γενικά είναι ικανοποιητική η εφαρμογή και ελοποίηση αυτού του προγράμματο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο η συζήτηση για την πολιτική συνοχής ε, και θεματικός στόχος, ε, προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλληψη των σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων. Άρθρα 9, παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης υπό την Επιτροπή Ρέτζη. Το λόγο έχει ο κύριος Σλοτόφσκι που είναι εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους κατέθεσαν τροπολογίες και τους ασκιώτες συζητητές για την πολύ καλή συνεργασία. Την περασμένη εβδομάδα συμφωνήσαμε επί του ε, συμβιβαστικού κειμένου που λαμβάνει υπόψη σχεδόν 30 εκ των 50 τροπολογιών ιδιαίτερε ευχαριστίε προ τον κύριο Μαρινέσκου που επέστησε την προσοχή μα στο γεγονό ότι ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε την ε, πρόταση σε ό,τι αφορά τα σημεία συμφόρηση ε, για τα βασικά και βοηθητικά δίκτυα. Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχή και το ΕΦΣΥ για προγράμματα όπως τα TNT και η άρση των σημείων συμφόρησης. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει ε, η Γενική Διεύθυνση MOVE να ε, εμπλακεί περισσότερο στην διαδικασία χάραξης πολιτικής και λήψη αποφάσεων ε, για τα προγράμματα χρηματοδότησης έργων υποδομών. Συμφωνώ τον κύριο Κράμερ για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις του και που μας υπενθύμησε την ανάγκη επανοικοδόμησης των διασυνεριακών ε, τμήματων υποδομών που ε, καταστράφησαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επεσήμανε επίση ότι είναι σημαντικό ε, να έχουμε υποδομές χρήσης ποδηλάτων και αυτές κάπως να συνδυάζονται με τους σιδηροδρόμους. Για να εξαλείψουμε τα σημεία συμφόρησης χρειάζομαστε όμως και χρηματοδοτικά μέσα. Ε, ζητείτε λοιπόν η απαραίτητη χρηματοδότηση για την περίοδο μετά το 2020. Και βεβαίω θα ήθελα να συζητήσω να στηρίξετε την νομοδότησή μου αύριο κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία ε, αλλά και στην Επιτροπή ΡΕΤΖΗ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Σχιώδης εισηγητές τώρα. Ο κύριος Βαντερκάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όπως ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος Σλοτόφσκι, και πάλι έχω την τιμή να αντικαθιστώ τον κύριο Μαρινέσκου και εξ ονόματός του μπορώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, για το έργο του και για την εκπόνηση του κειμένου. Είναι πολύ καλό που μετά από την ε, συζήτηση για το ΣΕΦ μπορούμε απευθείας να περάσουμε σε αυτό το θέμα το οποίο συνδέεται. Για έναν Πολωνό εισηγητή φαντάζομαι ότι δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να μπαίνει σε τέτοια χωράφια, αλλά νομίζω ότι ε, εκπώνησε μια γνωμοδότηση που είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη. Βέβαια και πάλι είναι ζήτημα η χρονική διάσταση. Όλα αυτά στην Ευρώπη παίρνουν πολύ χρόνο μέχρι να περάσουμε τελικά σε επενδύσεις. Και η λήψη αποφάσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρη στη δικασία και η υλοποίηση των αποφάσεων. Ε, νομίζω ότι η Επιτροπή Ρέτζι, ελπίζω μάλλον, να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μας, να συνεχίσουμε ε, στις επενδύσεις για τα δίκτυα TNT και μία παρατήρηση, εάν η Επιτροπή Ρέτζι δημιουργήσει νέα χόμπι, αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της Επιτροπής Μεταφορών. Γιατί έτσι χάνουμε τον στόχο μας. Και πάλι όμως ευχαριστούμε τον εισηγητή, πολύ ισορροπημένη γνωμοδότηση και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στις μελλοντικέ συζητήσεις. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστούμε τον κύριο Βαντερκάμπ. Ο Ισμαήλ Ερτούκ. Uh, Ευχαριστώ πολύ η ε, κυρία Γκραπίνη δεν μπορούσε να δώσει σήμερα, μου ζήτησε λοιπόν ε, να πάρω το λόγο. Και από πλευρά μας ευχαριστούμε τον εισηγητή. Πολύ σημαντική γνωμοδότηση εν ώψη και της ε, επερχόμενης πρότασης για το ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ. Θεωρούμε ότι πρέπει να ε, διατηρήσουμε και να εξυγχρονίσουμε τις υφιστάμενες υποδομές και νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικός τομός, ε, τομέας χρηματοδότησης και επενδύσεων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περαιτέρω χρηματοδότηση και αναφέρουμε ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν ε, οι διασυνοριακοί σύνδεσμοι που αυτή τη στιγμή μας λείπουν και τέλος, να σας πω ότι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες στηρίζουν ε, τους συμβιβασμού στους οποίους έχει καταλήξει ο εισηγητής. Ευχαριστούμε κύριε Ρτούκ. Ο κύριος Μίλτεμπιρχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγητή για το έργο του και την επικοδομητική του προσέγγιση και η ΆλΔε θα υποστηρίξει όλες τις συμβαστικές τροπολογίες και θα υπερψηφίσουμε ε, την πλειονότητα των τροπολογιών. Όμως θα θέλαμε να σταθούμε στην ουσία Τη νομοδότησης και θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες που είναι είτε ε, υπερβολικά συγκεκριμένε, είτε εκτός πεδίου εφαρμογή. Η τροπολογία 34 για παράδειγμα. Ε, για τι υποδομέ που έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Νομίζουμε ότι αυτό είναι πολύ περιοριστικό και συγκεκριμένο. Φυσικά και είναι κάτι το οποίο θα μα απασχολήσει στο μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία 2. Θα θέλαμε και εμεί αναθεώρηση των ε, πολιτικών συνοχή και όχι απλή αύξηση των κονδυλίων στο ε, ΠΔΠ. Είμαι συγκητή και για την έκθεση στη Ρέτζη, γι' αυτό θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμπεριλάβω τμήματα και αυτή τη γνωμοδότηση στην τελική έκθεση τη Ρέτζη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κράμαρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα τον εισηγητή. Όλος ιδιαίτερος. Δεν είναι και εύκολο να φτιάξει από τόσο πολλές τροπολογίες, τελικά 30 συμβαστικές, τις συμβαστικές τις βρήκα πολύ καλές. Και συμφωνήσαμε όλοι μάλιστα, εκτός από τον ε, Βαν Μίλτενμπερκ που θεωρεί ότι είναι υπερβολικά συγκεκριμένες διότι λείπουν, ε, δεν, πρέπει να αποκατασταθούν αυτοί οι λείποντες κρίκοι. Εδώ και 30 χρόνια όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε μια ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών δικτύων. Έχουμε δώσει δισεκατομμύρια που τελικώς οι χώρες μέλη τα διέθεσαν για δικά τους έργα και καμία προστιθέμενη αξία. Δηλαδή μένουμε σε, αυτή, σε αυτόν τον χωρισμό και όχι μόνο του Βερολίνου και της Γερμανίας αλλά όπλης της Ευρώπης. Μεταξύ Φράιμπουργκ και Κολμάρ καταστράφηκε η γέφυρα πάνω από το Ρήνο στον δεύτερο πόλεμο στα, από τα γερμανικά στρατεύματα και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί, ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Έχω και άλλα παραδείγματα στην πατρίδα σας, στην Ολλανδία. Και επί 30 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να κλείσουμε αυτά τα μικρά κενά. Δεν πρόκειται για ιδιαιτερότητες, πρόκειται για πράγματα αναγκαία για να αποκατασταθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αντιλαμβάνομαι αυτό που επιθυμείτε, να γίνουν ψηφοφορίε κατά τμήματα. Όμω, προ Θεού, έχουμε μια πλειοψηφία η οποία δεν θέλει να αγνοηθεί η ιστορία. Θέλουμε να ξεπεραστούν τα αποτελέσματά τη. Ήταν πολύ κακή υπόθεση η διαίρεση της Ευρώπης, αλλά θέλουμε να αποκατασταθεί η ενότητα. Δεύτερο που είναι σημαντικό για μένα. Έχουμε αυτή την υπόθεση τώρα με τις ε, κοινοπραξίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πέρασα μια φορά στην Ελβετία και μου είπαν εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, κοινοπραξίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και μου λέω μα γιατί μου λένε διότι τα κρίσιμα προβλήματα, οι ιδιώτες ούτως ή άλλως δεν βάζουν το χέρι στη τσέπη. Και όπου προκύπτει όφελος, καλύτερα να τα κάνουμε εμείς στο δημόσιο, δηλαδή να τα βάλει, να τα βάλει στη τσέπη του ιδιωτικού τομέα. Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν συμμετοχή όχι μόνο στις ζημίες αλλά και στα κέρδη και όχι να αναλαμβάνει το δημόσιο τις ζημίες ενώ τα κέρδη να τα κρατάει ο ιδιωτικός τομέας όπως έχει γίνει στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Γι' αυτό θέλουμε τουλάχιστον εδώ να υπάρξει πράγματι έντιμος και ισότιμος ανταγωνισμός και γι' αυτό παρακαλώ όλες και όλους να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Λάινερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λίγα σχόλια μόνο σχετικά με τις ε, συμβαστικές τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Η πρώτη μας παρατήρηση για την υπαριθμόν 2, όπου σημειώνεται ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα διαχειρίζονται διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής. Γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία η στενή συνεργασία των υπηρεσιών της Επιτροπής και νομίζω ότι έχουμε και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για να εξασφαλίζει το συντονισμό των προσπαθειών των υπηρεσιών μας. Δεν θεωρούμε ότι η εμπλοκή διαφόρων υπηρεσιών της Κομισιόν, Regio και άλλε θέτουν σε κίνδυνο την εναρμονισμένη προσέγγιση. Δεύτερο σχόλιο για τη συμβαστική τροπολογία 3 και θα επανέλθω σε μια παρατήρηση που κάναμε και στην τελευταία συνάντηση της ε, Επιτροπής σας για τον χαμηλό ρυθμό επιλογής ε, έργων και για το, για το Περιφερειακό Ταμείο, αλλά για τις μεταφορές έχουμε άνω του 60% και για επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών έχουμε ακόμα υψηλότερα ποσοστά ε, επιλογής μάλλον. Και για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη έχουμε ακόμα καλύτερο και για τα TNT έχουμε συντελεστή επιλογή στις τάξεις των 66%. Δεν θεωρούμε ότι είναι χαμηλή, χαμηλά τα ποσοστά αυτά επιλογής και σε ό,τι αφορά την συμβαστική 4, συμβαστική τροπολογία 4, όπου η Επιτροπή στα ζητεί από την Κομισιόν να κάνει ορισμένε αξιολογήσεις και να αναφέρει τα συμπεράσματα, επισημαίνω ότι έχουμε μηχανισμούς αξιολόγησης και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης των διευρωπαϊκών δικτύων. Έχουμε επίση μελέτες σε βάθος για μια ποικιλία θεμάτων μεταφορών αν προσθεθούν και άλλα κριτήρια, θα σημάνει αυτό μεγαλύτερη γεωγραφική επιβάρυνση των χωρών μελών. Και ειδικά για την εφαρμογή των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, αυτά είναι διαφανή και είναι βεβαίως διαθέσιμα στο 10T Tool, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της Επιτροπής σας και βεβαίως και το κοινό. Αυτά είναι τα, τα σχόλια που ήθελα να κάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Λάιρε innego, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και να σας καλέσω να υπερψηφίσετε την έκθεση αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο λοιπόν έχουμε την ψηφοφορία στις 9 το πρωί και θα κλείσω τώρα την συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα ξαναρχίσουμε στις 5.30 μόνο με τους συντονιστέ και κλεισμένων των θυρών στις 5.30. Τους υπόλοιπους θα τους ξαναδώ αύριο.